Κύριοι, συνάδελφοι, παρακαλώ να περάσουμε στο σημείο 8 της ημερήσιας ε, διάταξης, έκθεση Τάνοκ για το Μαυροβούνιο. Κύριε Τάνοκ, έχετε να πείτε κάτι. Όχι κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Τα είπαμε χθε και με τους Κιώδης όπου αποφάνθηκαν και εκείνοι. Εκτός από την ομάδα Γκουε όλοι ε, υποστήριξαν τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Οπότε είναι αυτά τα οποία έχουμε ψηφίσει με μεγάλη πλειοψηφία. Ευχαριστώ. Αρχίζουμε λοιπόν συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ε, τροπολογία 10, ε, δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Συμβιβαστική 2, 2, υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 15, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 20 υπέρ κατά αποχές έλεγχος νομίζω ότι έχει γίνει δεκτή ich habe die Zeit. Good morning. It was, on, it was early, but only for Silvio. Der schnelle Italiener hat die Stoppuhr angestellt gehabt. Νομίζω ότι ο ταχύτατος Ιταλός είχε βάλει το χρονόμετρο. Πέρασε της ψηφοφορίας. 26 υπέρ 24 κατά δεκτή. 21 υπέρ κατά αποχές νομίζω δεκτή με την ίδια πλειοψηφία έλεγχος 21. την 21 ψηφίζουμε <laughs> Ja, aber ihr habt anders abgestimmt. Okay, geschlossen? Ja. Ψηφίσατε διαφορετικά όμως, λέει ο πρόεδρος πέρασε το ΕΛΚ στην ώρα της αλήθειας σε σαφές ναι, υπέρ, οπότε δεκτό. 22, υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Πέρασε. 26 προς 25 δεκτή 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος την 30 ψηφίζουμε 30, 30 24 υπέρ, 22 κατά δεκτή 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή 32 υπέρ κατά αποχές έλεγχος στην 32 είμαστε πέρας 23 υπέρ 26 κατά απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος ζητείται Die Abstimmung ist geschlossen. Πέρας. 23 προς 28 απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. 35 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Die Abstimmung ist geschlossen. Πέρας ψηφοφορίας. 29, υπέρ 22 κατά δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 38. 38 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ. 42 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 43 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τώρα θα ψηφίσουμε την 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 53 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές φαίνεται να γίνεται δεκτό 56 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή η 60 τώρα μόνο το δεύτερο τμήμα. Στην 60 είμαστε. Μόνο το δεύτερο τμήμα, μάλιστα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ψήφισαν κατά οι φιλελεύθεροι. Ναι, απερίφθη, απερίφθη, ναι. Ψήφισαν κατά. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τμήμα 1 της 70 υπέρ κατά αποχές δεκτό 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές δεκτή 74 υπέρ να κάνω ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 73 την 73 η 69 απορρίφθηκε η 73. Η δεκτή. Δεν είναι. Δεν με, δεν με πιστεύετε. Πέρας. Δεκτή. Με σαφή πλειοψηφία. 74 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. Απορρίφθηκε λέτε. 75 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 76 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 79 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 80 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 81 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 82 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 83 υπέρ, κατά δεκτή 84 υπέρ κατά οι φιλελεύθεροι πώς εψήφισαν είπαν ναι δεκτή λοιπόν 85 υπέρ κατά αποχές δεκτή 86 υπέρ κατά αποχές δεκτή 87 υπέρ κατά αποχές δεκτή 88 υπέρ κατά αποχές δεκτή 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ενενήντα υπέρ κατά αποχές δεκτή 91 υπέρ κατά αποχές δεκτή 92 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή Ποιος είναι υπέρ... Όχι, ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε τώρα επί του συνόλου. Πέρας. Πενήντα υπέρ, μία ψήφος κατά Κύριε Τάνοξ, σας υπόσχομαι να τον βρούμε αυτόν τον ένα. Λοιπόν, έκθεση Κοβάλ, σχέδιο γνωμοδότησης. Μία ηλεκτρονική ψηφοφορία πρέπει να γίνει. Κύριε Κόβαλ, έχετε να πείτε τίποτα. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Ποιος είναι αυτός. Συνάδελφοι, προχωρούμε στην έκθεση για την Κροατία. Ο εισηγητής, ε, ο κύριος Ρούτσεκ, είναι πρώτη ανταλλαγή απόψεων εδώ, επί της εκθέσεως και μάλλον πρόκειται για την τελευταία έκθεση που αφορά την διεύρυνση προς τη χώρα αυτή. Η Κροατία την 1η Ιουλίου του 2013 πρόκειται να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 20 κράτη-μέλη και η Κροατία, 21, α, 21 εντωμεταξύ, έχουν κυρώσει την ε, συνθήκη προσχώρησης. Περιμένουμε σε εύθετο χρόνο να προχωρήσουν και οι άλλες χώρες στην κύρωση και ελπίζουμε τους επόμενους μήνες η Κροατία να διευθετήσει αυτά τα δέκα καθήκοντα, τις δέκα συγκεκριμένες ενέργειες όπως αναφέρει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Οκτωβρίου. Την τελευταία έκθεση παρακολούθησης θα τη δούμε το Μάρτιο. Οπότε όταν πληρούμε και εμείς και η Κροατία τις προϋποθέσεις θα μπορέσει να τηρηθεί η ημερομηνία της 1ης Ιουλίου. Αυτό αν ε, λειτουργούσε θα ήταν ευπρόσδεκτο. Συνάδελφε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ήδη αναφέρατε κι εσείς Πρόεδρε, είναι η τελευταία έκθεση πρόοδου που συζητάμε για την Κροατία εφόσον όλα πάνε καλά, που ελπίζω και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Τον Ιούλιο του 2013 η Κροατία θα γίνει το 28ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να συγχαρώ λοιπόν τους Κροάτες συναδέρφους και ολόκληρη την Κροατία, γιατί για την Κροατία αποτελεί ένα ιστορική σημασία ε, επίτευγμα, η πρόοδος που έχει πετύχει η χώρα. Είναι λοιπόν ένα επίτευγμα, μια πρόοδος για ολόκληρη την πολιτική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια από τις πιο επιτυχείς πολιτικές μας. Το σχέδιο έκθεσης περνάει τρία κυρίως μηνύματα. Πρώτα απ' όλα το ότι η Κροατία έχει μπει στο δρόμο προκειμένου να αποτελέσει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούλιο. Το Ζάκρεπ έχει πετύχει όλους τους στόχους που αναφέρει η έκθεση της Επιτροπής. Υπάρχουν δύο στόχοι που μένουν. Μίλησα με τον Αντιπρόεδρο Μίμητσα ο οποίος υποσχέθηκε ότι τον Μάρτιο θα έχουν επιτευχθεί και αυτοί οι δύο στόχοι. Και πρόκειται για την ιδιωτικοποίηση ενός ναυπηγείου που παραμένει και τις διευκολύνσεις στην Αδριατική ακτή ανάμεσα στην Κροατία και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Πώς γίνεται το πέρασμα δηλαδή των συνόρων εκεί. Η Κροατία λοιπόν είναι μια όρημη δημοκρατία. Έχει κοινωνική οικονομία, έχει αναλάβει τις υποχρώσεις της ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στην έκθεσή μου ζητάω από τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμα επικυρώσει την συνθήκη προσχώρησης να το κάνουν αυτό. 21 χώρες η Γαλλία είναι τελευταία που επικύρωσε την συνθήκη αυτή προσχώρησης. Έχουν ήδη επικυρώσει. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την επικύρωση όσον αφορά τη Σλοβενία. Κατά σύμπτωση σήμερα οι ειδικοί οικονομικοί πυρογνώμονες και από την Κροατία και από την Σλοβενία συναντιούνται και θα συζητήσουν για άλλη μια φορά αυτό το ακαθόβες θέμα της Βλάσκα Μπάνκα. Ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση σε αυτό και έτσι και η Σλοβενία να μπορέσει τελικά να επικυρώσει τη συνθήκη αυτή προσχώρησης. Δεύτερον, η έκθεσή μου υπογραμμίζει το βιώσιμο των μεταρρυθμίσεων μετά την ε, προσχώρηση προκειμένου οι πολίτες της Κροατίας να μπορέσουν να αποφεληθούν πλήρως από την προσχώρηση αυτή. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με το κράτος δικαίου μια που υπάρχει περιθώριο δελτίωσης προκειμένου να ενισχυθούν οι θεσμοί της χώρας, η ανεξαρτησία της ε, δικαιοσύνης, ε, νόμοι και δίωξη κατά της διαφθοράς και τέλος το θέμα της δημόσιας δίκησης. Τι χρειάζεται τώρα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που χρειάζεται είναι ε, το ΣΑΜΠΟΡ που είναι το κρατικό κοινοβούλιο να έχει την εποπτεία όλων αυτών και έτσι να μπορέσει να βοηθήσει τις εξελίξεις στην κοινωνία. Και οι πολιτικοί που περνάνε τους νόμους να λογοδοτούν μετά στον κόσμο. Η έκθεσή μου επίσης αναφέρεται πολύ στις επιπτώσεις στην ε, γύρω περιοχή. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε λοιπόν είναι να ενθαρρύνουμε την Κροατία να αναλάβει ενεργό ρόλο προκειμένου να εφαρμοστούν οι ευρωπαϊκές πολιτικές στην περιοχή και για την ε, διεύρυνση, για τις ευρωπαϊκές αξίες γενικότερα. Και είναι πολύ καλό να μπορέσει να μοιραστεί με τους γείτονές της την εμπειρία της από όλη τη διαδικασία αυτή που οδηγεί στην ε, προσχώρησή της. Ο ρόλος που βλέπω εγώ για την Κροατία είναι ότι η Κροατία πρέπει να είναι δραστήρια να αντιμετωπίσει τα διμερεί ζητήματα που τίθενται με τις γείτονες χώρες, ώστε κάποιες ενδυνάμει διαμάχες να μην εμποδίζουν την ε, διαδικασία προσχώρησης. Η Κροατία δηλαδή μπορεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στα Βαλκάνια, να αποτελέσει το μοντέλο αλλά και την κινητήριο δύναμη για παρετέρω διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρετέρω προσχωρήσεις χωρών, το Μαυροβούνι για παράδειγμα, που ήδη συζητήσαμε χτες. Συνεπώ, αγαπητοί συνάδελφοι, περιμένω τώρα τα δικά σας τα σχόλια. Θα υπάρξουν βέβαια κάποιε τροπολογίε. Σε δύο εβδομάδε στο Στρασβούργο μπορούμε να συζητήσουμε τις τροπολογίες αυτές και έτσι να έχουμε μια καλή έκθεση και να συνεισφέρουμε με αυτόν τον τρόπο στην επιτυχία της προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μπέρντ Πόσελ από το ΕΛΚ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Ε, είπατε ότι ε, δεν μπορεί κανείς να, παρά να με δει. Και εσείς το ίδιο θα έλεγα. Ευχαριστώ τον κύριο Ρούτσερ για την εξαιρετική έκθεση, την εξαιρετική δουλειά, την άριστη συνεργασία με τους Σκιώδης. Υπάρχει ευρεία και σε βάθος συμφωνία εδώ. Πρέπει όμως να πω ότι πρέπει να αναδείξουμε κάποια θέματα, να, δώσουμε, να βάλουμε κάποιες προτεραιότητες. Μία προτεραιότητα είναι η αναγνώριση των τωρινών προσπαθειών της κροατικής κυβέρνησης, ιδιαίτερα του Αντιπροέδρου Μίμητσα που τον ξέρουμε όλοι καλά και ε, θέλει να διαφυλάξει τη συνοχή ε, και τις μεταρρυθμίσεις. Από την Κροατία κάποιες άλλες χώρες στην περιοχή μπορούν να εντλήσουν διδάγματα διότι αυτή η προσέγγιση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι θέμα κομματικής πολιτικής, είναι ένα θέμα διαπαραταξιακό. Ε, θα πρέπει να γίνει με συνένεση. Αυτό γίνεται στην Κροατία και πρέπει να πω ότι είμαι πεπισμένος ότι μέχρι το Μάρτιο το αργότερο η χώρα αυτή θα έχει κλείσει τα θέματα που υπολείπονται, τα δέκα αυτά και κατά τα άλλα έχουμε συμφωνήσει με την προσχώρηση. Δεύτερον, πρέπει να ασκήσουμε όλοι μαζί πιέσεις για τη διαδικασία κύρωσης. Χαίρομαι γιατί η Γαλλία, μία από τις μεγάλες χώρες που δεν είχαν κυρώσει τη συνθήκη, προχώρησαν στην κύρωση, όμως ε, διατυπώνω την δυσαρέσκειά μου για τη δική μου τη χώρα, τη Γερμανία, και απευθύνω έκκληση και στην καγκελάριο να προχωρήσει. Σήμερα είναι η επέτειο τη συμφωνία συνθήκη των Ηλυσίων και καλό θα ήταν και η Γερμανία όπω η Γαλλία να προχωρήσει στην κύρωση, ούτω ώστε να είμαστε έτοιμοι μέχρι την 1η Ιουλίου και να μην είναι αυτό αφορμή για καθυστέρηση. Τρίτο. Να συμπληρώσουμε προσθέτοντας την έκθεση, προσθέτοντας ένα εδάφιο για να αναφέρομαι την εξαιρετική συνεργασία με τους συναδέλφους από την Κροατία οι παρατηρητές, ε, ε, τους παρατηρητές από την Κροατία που ε, συνεργάζονται εξαιρετικά και θα πρέπει να αναλάβουν ενεργό δράση το αργότερο την 1η Ιουλίου. Τελευταίο θέμα που νομίζω ότι είναι επίσης σημαντικό και πρέπει να προσεχτεί οι προετοιμασίες για την διαδικασία προσχώρησης δεν θα πρέπει να πέσουν θύμα εθνικών εκλογών και προεκλογικών εκστρατιών και απευθύνομαι εδώ συγκεκριμένα στους Σλοβαίνους συναδέλφους. Υπάρχει πάλι κυβερνητική κρίση στη Σλοβενία με πολλές αναταραχές στην εσωτερική πολιτική, βίες αναταραχές και εκφράζω την ελπίδα προβλήματα ε, γειτονίας να μην θεματοποιούνται με τρόπο τέτοιο ούτως ώστε να έχουμε ε, μπλοκάρισμα της διαδικασίας. Εγώ έχω ασχοληθεί με τη χώρα, ήμουν εισηγητής για τη Σλοβενία και την υποστήριξα πολλές φορές πολύ, αλλά παρακαλώ να φροντίσει η Σλοβενία εν προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις. Ευχαριστώ, συναδελφέ. Ναι, και εγώ το τελευταίο κομμάτι της έκκλησης το υποστηρίζω και υποστηρίζω και αυτό που είπατε για τη χώρα μας. Ο κύριος Κασίν, παρακαλώ. <coughs> Σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, καταρχήν επιτρέψατε μου να συγχαρώ τον κύριο Ρότσεκ για μια εξαιρετική, ισορροπημένη και πολύ θετική έκθεση. Η Κροατία όντως χρειάζεται ενθάρρυνση για να μπορέσει να ολοκληρώσει τα... τις εργασίες σε το χρόνο, να βελτιώσει την αυτοπεποίθησή της έτσι και να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα όλο ιδιαίτερος να επενέσω την ε, δουλειά που έχει γίνει όσον αφορά την ε, βελτίωση των σχέσεων ε, της καλής γειτονίας. Τελευταία επίσκεψη δε του Προέδρου Μιλάνοβιτς στην Σερβία ήταν μια πολύ καλή, ένα πολύ μια πολύ καλή ε, πρωτοβουλία ε, και μάλιστα να σας πω ότι και εμείς θέλουμε να ενθαρρύνουμε την Κροατία, όμως ε, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, άρα η διαδικασία επικύρωσης δεν θα ξεκινήσει. Αυτό δεν έχει να κάνει με την κυβερνητική κρίση. Η σχέση μας με την Κροατία είναι στρατηγική σημασία στη Σλοβενία και άσχετα από την κυβέρνηση που έχουμε, οι στρατηγικές προτεραιότητες παραμένουν σταθερές και δεν υπάρχει αμφιβολία για όλα αυτά. Αλλά φυσικά πρέπει σαφώς να πούμε ποιος είναι, ποιο είναι το ζουμί αυτής της υπόθεσης. Αυτά που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής δεν γίνονται τηρητά. Δεν τηρούνται, με συγχωρείτε. Η κροατική νομοθεσία όπως και η δική μας, βασίζονται στο pacta sunt servanta Ότι δηλαδή οι υποχρεώσεις που έχουν αναλυφθεί πρέπει να ε, υλοποιηθούν. Εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επικύρωση. Ο συνάδελφος Πόσελτ ανέφερε ως οι δυο εθνικοί εμπειρογνώμονες για την υπόθεση της ε, Τράπεζας Λουμπλιάνα συναντώνται, αλλά δεν πρόκειται να λυθεί το ζήτημα γιατί δεν έχουν προτείνει μάλλον, έχουν προτείνει να διωχθεί ποινικά η τράπεζα, η, τράπε, η κυβέρνηση το έκανε, αλλά ακόμα δεν έχει ληφθεί η ε, δικαστική απόφαση. Να αναφέρω δε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός Αντρόποβιτς είπε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μιλάνο στο Βελιγράδι πως θα ήταν πιο επικοδομητικό και παραγωγικό να συναντώνταν οι πρωθυπουργοί Σλοβενίας με Κροατία για να λυθούν τα προβλήματα τα κράτη-μέλη μας είναι κυρίαρχα και δεν μπορώ να σκεφτώ ούτε έναν βουλευτή του Εθνικού μας Κοινοβουλίου που θα υπερψήφιζε την επικύρωση εάν δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες. Οι συγκινησιακές προσεγγίσεις δεν είναι ε, σκόπιμες αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει λογικά να σκεφτούμε. Πιστεύω λοιπόν πως έχουμε ακόμα χρόνο, πρέπει να ε, είμαστε λογικοί και ψύχρεμοι και είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά θα ολοκληρωθούν σε αυτό το χρόνο προς όφελος της Κροατίας, της περιοχής και της Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ρούτσεκ, τον εισηγητή μας, για το σχέδιο έκθεσης που παρουσιάζει. Ωραία είναι που είναι η τελευταία φορά που η Επιτροπή μας ασχολείται με την Κροατία ως υποψήφια χώρα. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Αλλά από την άλλη, Γίτσε λέει σε κάποιον που φτερνίστηκε ομιλήτρια. Ε, από την άλλη μεριά λοιπόν πρέπει να προσέχουμε τι ακριβώς γίνεται. Η Κροατία έχει σίγουρα δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Παραμένουν όμως ακόμα κάποια ζητήματα. Και δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματα να προχωρήσουν πολύ γρήγορα. Πρέπει να επιμείνουμε να γίνει δουλειά που πρέπει να γίνει. Και γι' αυτό θέλω να αναφερθώ στο ένα θέμα που είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, εδώ μένουν αρκετά πράγματα να γίνουν. Η κυβέρνηση της Κροατίας πρέπει πιο αποφασιστικά να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να φροντίσει λίγο και για το θέμα της δημόσιας δίκησης, να λογοδοτεί περισσότερο η δίκηση απέναντι στον κόσμο. Και εδώ σας παραπέμπω στην σύσταση του Λεκτικού Συνεδρίου που αναφέρθηκε στη διαχείριση του Ταμείου Συνοχής και ότι θα έπρεπε να υπάρξει κάποια αναβάθμιση της ικανότητας της κρατικής δίκησης. Βλέπετε, αναρωτιόμαστε πάντα πού πάνε τα χρήματα. Δεν θα έπρεπε και εδώ να έχουμε μια κατάσταση που, με το, που θα αναγκαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει τη χρηματοδότηση επειδή θα διαπιστώσει ότι δεν γίνεται σωστή διαχείριση. Το τελευταίο είναι το θέμα των εγκλημάτων πολέμου. Εδώ πρέπει επίσης να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία συμφιλίωσης. Πάντως από πλευρά της Κροατίας πρέπει να το δούμε και αλλιώς. Να δούμε τι κάνουν οι δικές μας οι χώρες. Αναφερθήκατε στη Γερμανία. Να σας πω ότι ο κύριος Λάμαρτ, πρόεδρος της Bundestag, έχει αφισβητήσει την προσχώρηση της Κροατίας, κάτι το οποίο εγώ βρήκα ότι είναι ιδιαίτερα ατυχές. Θέλω να πω λοιπόν στους συναδέλφους από το κόμμα αυτό να το φροντίσουν. Δεν είναι το δικό μου το κόμμα που μπλοκάρει την ε, υπογραφή αυτή, την κύρωση. Έπειτα, να μην ε, δεχτούμε ε, μέτρα προσωρινά, παρά μόνο όταν είναι εντελώς αναγκαίο. Για την ελεύθερη κυκλοφορία, για παράδειγμα, μόνο σε έσχατη περίπτωση να δεχτούμε τον περιορισμό αυτό, μόνο αν όντω διαπιστώνουμε ότι θα υπάρξει στρέβλωση στην αγορά. Και το τελευταίο, το μάθημα δηλαδή που πρέπει να πάρουμε από τη διαδικασία προσχώρησης της Κροατίας εν ώψη επόμενων ε, προσχωρήσεων, είναι το ότι η διαδικασία έχει γίνει πιο διάφανη αλλά θα πρέπει περισσότερο ακόμα να συμμετέχει το κοινοβούλιο της κάθε χώρας και η κοινωνία των πολιτών. Σίγουρα ήταν επιτυχία η διαδικασία μέχρι τώρα και νομιμοποιεί ακόμα περισσότερο τη διαδικασία. Στηρίζουμε την διεύρυνση αυτή και από τις δύο πλευρές. Από εκεί και πέρα με τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές είχαμε πολύ καλές συζητήσεις και όντως ελπίζω και εγώ να είναι τελευταία φορά που ασχολούμαστε με την Κροατία ως υποψήφια χώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να πω ότι ο πρόεδρος Λάμερ δεν θέλει να μπλοκάρει τίποτε, απλώς είπε ότι η Κροατία θα πρέπει να ασχοληθεί με τις 10 προτάσεις και συγκεκριμένες ενέργειες που προσδιορίσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι αυτό είναι σημαντικό για να κρίνουμε την κύρωση. Τίποτε δεν παρεμποδίζεται και λέω ότι απλώς όταν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις που πρέπει να υλοποιηθούν, ε, θα πρέπει να υλοποιηθούν για να ε, σεβαστούν τους κανόνες που έχουν τεθεί. Ο κύριος Στάνοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ε, ομάδα μας η ECR είναι υπέρ της διεύρυνσης και της προσχώρησης ε, της Κροατίας. Συμφωνώ με την κυρία Μπράντερ για το κράτος δικαίου, τη διαφθορά και την καταπολέμησή τους. Αυτό σημαίνει συνεχιζόμενη μάχη όχι μόνο στις υποψήφιες χώρες αλλά και σε κάποια κράτη-μέλη μας. Έχουμε ε, μάθει από προηγούμενες ε, διευρύνσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυστηρότερη τώρα και καλά κάνει. Και βέβαια συγχαίρω τον εισηγητή για την καλή του δουλειά, τον κύριο Ρούτσεκ. Ε, ένας όρος που δεν έχει συζητηθεί, μια ανησυχία μου, και αυτό είναι θέμα που με αφορά γιατί είμαι εισηγητή για το Μαυροβούνιο, και ιδιαίτερα στο φως της εκστρατείας της Σλοβενίας και τις προηγούμενες προσπάθειες και τις διμερείς διαφορές για τα σύνορα που ήταν αντικείμενο δημοψηφίσματος και κόντεψε να εμποδίσει τελείω την προσχώρηση της Κροατίας. Νομίζω υπάρχει θέμα εδαφικό μεταξύ Κροατίας και Μαυροβουνίου και έμαθα και ανησύχησα πρόσφατα ότι το θέμα δεν λύθηκε. Νόμιζα ότι είχε λυθεί στο Διεθνές Δικαστήριο, φαίνεται όμως ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο και ανησυχώ όταν θα γίνει κράτος μέλος η Κροατία, φοβάμαι μην ε, χρησιμοποιήσει την ιδιότητά της ως μέλους για να αποκλείσει το ε, Μαυροβούνιο λόγω διμερούς διαφοράς, ε, γιατί ο πρώτος που θα προσχωρήσει ε, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στους επόμενους σε σχέση με πολιετής διαφορές. Ανησυχούμε λοιπόν ότι μπορεί η Κροατία να αξιοποιήσει την ιδιότητα του κράτους μέλους για να ε, δημιουργήσει πρόβλημα λόγω διμερών διαφορών με τη Σερβία. Τι διασφαλίσεις έχουμε λοιπόν από την κροατική κυβέρνηση ότι δεν θα επιτρέψουν την ε, ένταξη για να μπλοκάρουν την ε, προσχώρηση αργότερα και του Μαυροβουνίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ τον κύριο Ρούτσεκ για την δουλειά που έχει κάνει πάνω στην έκθεση αυτή. Και κυρίως γιατί έχει αντιμετωπίσει το θέμα πολύ επικοδομητικά, με πολύ σωστή προσέγγιση. Η Κροατία με αυτόν τον τρόπο θα γίνει πλήρες μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα υπάρχουν διάφορα θέματα που εξακολουθούν βέβαια να τίθεται. Πρώτα απ' όλα, η αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης. Είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να γίνει δουλειά. Όμως η Κροατία πρέπει να εφαρμόσει πρώτα απ' όλα να ολοκληρώσει και να εφαρμόσει την στρατηγική για το δικαστικό της σώμα. Να καταπολεμήσει την διαφθορά, επίσης είπαμε. Έπειτα η κυβέρνηση πρέπει να ασχοληθεί με ένα νέο πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς και να γίνουν οι έρευνες που έχουν αποφασιστεί για την υγεία. Χρειάζεται πάντως περισσότερη αποτελεσματικότητα για να καταπολεμηθεί η τοπική διαφθορά και η διαφθορά στον τομέα των ε, δημοσίων ε, συμβάσεων. Επίσης πρέπει να ενισχυθεί το σύστημα για να μην υπάρχει ε, σύγκρουση συμφερόντων. Είναι ζωτική σημασία σε αυτά. Θέλω επίσης να σας πω ότι ο ρόλος της Κροατίας στην ε, περιφερειακή συνεργασία είναι ιδιαίτερα θετικός. Και γι' αυτό θέλω όλους ιδιαίτερος να αναφερθώ εδώ στα βήματα που έχουν γίνει για τις σχέσεις με τη Σερβία. Παρ' όλα αυτά πρέπει να γίνει ακόμα πρόοδος όσον αφορά το διασυνοριακό, τη διασυνοριακή διάβαση του διαδρόμου του νέου για να λυθούν και αυτά τα προβλήματα με του, τις γείτονες χώρες. Ελπίζω ότι σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να υποδεχτούμε επίσημα την Κροατία ως ε, πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την 1η Ιουλίου να γίνει αυτό. Πάντως, να πω στην Κροατία ότι με το που θα γίνουν πλήρη μέλη δεν σταματάει δουλειά, πρέπει να συνεχίσουν να δουλεύουν σκληρά έτσι ώστε να διαλυθούν ό,τι τελευταίες αμφιβολίες μπορεί να υπάρχουν ακόμα στα μυαλά ορισμένων για το κατά πόσο είναι κατάλληλη στιγμή ή όχι να δεχτούμε την Κροατία ως πλήρες μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι θέμα εθνικής υπερηφάνειας, πιστεύω, και η Κροατία μπορεί να το πετύχει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αγκουράκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι από όλη αυτή τη διαδικασία ε, για την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο τελευταίο στάδιο της πραγματικά ε, και από την έκθεση που συζητάμε σήμερα φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Αλλιώ δεν μπορώ να, ε, για το λαό της Κροατίας θέλω να πω και οι συνέπειε είναι πάρα πολύ βαριές για τους εργαζομένους δεν μπορώ διαφορετικά να, να ερμηνεύσω το σημείο 13 της έκθεσης, η οποία, το οποίο ε, σημείο 13 ενθαρρύνει την Κροατία να πραγματοποιήσει και άλλες διαθροτικές μεταρρυθμίσεις, που σημαίνει ε, ιδιωτικοποίηση, που σημαίνει ανεργία, που σημαίνει φτώχεια και που σημαίνει, αν θέλετε, και μετανάστευση. Και θα ήθελα μια απάντηση από τον κύριο εισηγητή για το θέμα των ναυπηγείων, για την ιδιωτικοποίησή του. Ξέρω ότι είναι ένα τεράστιο θέμα, γιατί είναι χιλιάδε οι θέσει εργασία οι οποίε θα χαθούν και δεν υπάρχει εναλλακτικό πρόγραμμα, όπω δεν υπάρχει και πουθενά. Δεύτερο ζήτημα είναι για τις λεγόμενες διμερείς ε, διαφορές. Από ό,τι βλέπετε κύριε Πρόεδρε η διαδικασία ένταξης δεν είχε οδηγήσει σε μια άλλη θεώρηση ε, προβλημάτων του διεθνού δικαίου. Για μένα τα ζητήματα των συνόρων δεν είναι ζητήματα διμερών σχέσεων, είναι ζητήματα διεθνών σχέσεων και υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, κατά την άποψή μου, το ότι υπάρχουν ανοιχτά τέτοια ζητήματα τη στιγμή που και η Κροατία και το Μαυροβούνιο είναι μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σέβονται το διεθνέ δίκαιο και ακόμα δεν έχουν μπορέσει να λύσουν αυτό το πρόβλημα ε, δεν ξέρω τι γίνεται και με το θέμα με την Σλοβενία, με τα θαλάσσια σύνορα ε, που υπήρχαν. Τρίτο ζήτημα, με ανησυχεί ιδιαίτερα η αναφορά στο θέμα της συμφιλίωσης, στο σημείο 18, ε, όμως ε, ε, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τα Εγκλήματα της Ιουκοσλαβίας και γενικά το διεθνές πλαίσιο δεν βοηθάει στην συμφιλίωση των λαών στα Βαλκάνια με τις συγκεκριμένε αποφάσεις που έχουν επαρθεί στο παρελθόν. Τελευταία, θα ήθελα μια μεγαλύτερη επιμονή ε, εκ μέρους των κροατικών αρχών στο θέμα των μετατοπισμένων και στο θέμα των ε, προσφύγων. Η έκθεση κάτι πάει να πει, θα ήθελα περισσότερα στοιχεία γιατί πραγματικά είναι ένα τεράστιο ζήτημα ε, που δεν έχει λυθεί ακόμα και εφόσον δεν θα λυθεί θα υπάρχουν προβλήματα στο μέλλον. Τέλος, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν πιο συγκεκριμένες διατυπώσεις. Παραδείγματος χάρη πάλι θα αναφερθώ στο θέμα στο, στο σημείο 21 της έκθεσης όπου γίνεται λόγος για διμερείς διαφορές χωρίς η έκθεση να τις προσδιορίζει περισσότερο. Και όταν μιλάμε για τέτοια σοβαρά κείμενα νομίζω θα έπρεπε να είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Με όλα αυτά ε, το κόμμα μου και εγώ προσωπικά εξακολουθώ να, είμαι αντίθετος με την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς γιατί θεωρώ ότι οι συνέπειες του εργαζόμενων θα είναι πολύ χειρότερες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. 20 χρόνια μετά την ε, αναγνώριση, 13 χρόνια μετά από θεσμικούς θεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 8 χρόνια σχεδόν από τότε που άρχισαν οι διαπραγματεύσεις, η δημοκρατία της Κροατίας φτάνει στον κύριο στόχο της. Το πλήρες μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πέρα από οποιοδήποτε πολιτικό στόχο, αποτελεί ένα πολύπλευρο στόχο, όχι μόνο της κυβέρνησης, αλλά και των επιχειρηματιών, της κοινωνίας των πολιτών, των συνδικάτων, αλλά και των ατόμων, των πολιτών. Ήταν η πρώτη χώρα που ζήτησε προσχώρηση η Κροατία τον 21ο αιώνα και είναι η πρώτη χώρα η οποία επηρεάστηκε τόσο πολύ από τον πόλεμο στην ε, τέως Γιουγκοσλοβία και ζήτησε προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει εμπειρία δηλαδή από τον πόλεμο εκεί, αντιμετώπισε δύσκολες καταστάσεις και δύσκολα κριτήρια προκειμένου να μπορέσει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για χρόνια η Κροατία ε, αναδιαρθρώθηκε προς το καλύτερο και προς όφελος των πολιτών της. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να στηρίξουμε ε, τι γείτονες χώρες να προχωρήσουν και αυτοί στις ίδιες διαδικασίες και να μην μπλοκάρουμε ε, λόγω διμερών διαφορών την προσχώρησή τους. Η κυβέρνησή μας αυτά τα έχει πει ξεκάθαρα. Ναι, είμαστε κοντά στον ε, στόχο μας αυτό για να γίνουμε μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα. Τα λέει αυτά η έκθεση εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Οκτώβριο που μας πέρασε όπου αναφέρονται οι στόχοι που έχουμε πετύχει, αλλά και ποιε είναι οι τελευταίε προσπάθειε που μένει ακόμα να γίνουν. Η κυβέρνηση τη Κροατία πήρε πολύ σοβαρά την έκθεση αυτή. Όσον αφορά την ολοκλήρωση των 10 στόχων, έχουν περίπου γίνει. Και η δουλειά θα έχει γίνει πριν τα τέλη Μαρτίου πλήρω με ίσω μία μόνο εξαίρεση. Η έκθεση λέει ότι 21 χώρες μέλη έχουν ήδη κυρώσει την συνθήκη προσχώρησης. Ε, Μάλιστα η Γαλλία την προηγούμενη εβδομάδα ε, κύρωσε τη συμφωνία αυτή και η Βουλή των Λόρδων την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε, πιστεύω και η Γερμανία ότι θα το κάνει, και οι υπόλοιπε χώρες μέσα στο Φεβρουάριο. Έτσι ο αριθμός κύρωσης θα είναι πολύ υψηλότερο στη στιγμή που θα κλεθούμε να εγκρίνουμε αυτή την έκθεση, να την ψηφίσουμε. Η έκθεση είναι πάρα πολύ καλή και συμπεριλαμβάνει όλες τις πτυχές. Θέλω γι' αυτό να συγχαρώ τον εισηγητή και να θυμίσω ότι η τελευταία έκθεση εποπτείας της Επιτροπής θα παρουσιαστεί τον Μάρτιο του 2013. Κύριε Σόπφλη, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στον Λίμπο Ρούτσεκ για την πολύ καλή περιεκτική έκθεση. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που ακούσαμε. Ίσως όμως δεν είμαι τόσο αισιόδοξο όσο οι περισσότεροι σε σχέση με την 1η Ιουλίου. Ελπίζω να αποδειχθώ λάθος, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και εσωτερικά και διεθνή ε, προσκόμματα και διμερεί θέματα και θέματα κύρωσης. Ελπίζω να αποδειχθώ ότι κάνω λάθος, να αποδειχθεί ότι κάνω λάθος. Τι θα κάνουμε όμως αν δεν τηρηθεί η ημερομηνία της 1ης Ιουλίου. Δεν πρέπει να έχουμε έναν οδικό χάρτη, να δούμε τις επιπτώσεις, να είμαστε έτοιμοι, όχι μόνο για την Κροατία, αλλά για όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Θα υπάρξουν επιπτώσεις αν ε, πάει προς πίσω η ημερομηνία πάει για το τέλος του έτους, νομίζω ότι θα υπάρξει μεγάλη απογοήτευση, μπορεί οι τμήματα της κοινή γνώμης να ταχθούν κατά περαιτέρω διευρύνσεων. Ελπίζω λοιπόν να αποδειχθεί ότι κάνω λάθος, αλλά αν υπάρξει καθυστέρηση πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουν. Ευχαριστώ. Η κυρία... Ό, όχι, όχι, πρώτα ο κύριος ο Σπόσελτ πριν από την Επίτροπη. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αλλά θέλω να αναφέρω κάποια στοιχεία. Ήδη ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίσαμε επίσημα και δεσμευτικά για την, ε, για την προσχώρηση. Κάνουμε κάποιες διορθώσεις, αλλά υπάρχει η δέσμευσή μας. Επίσης, ο κομμουνιστής ε, συνάδελφος ε, θέλει να προστατέψει τους Κροάτες εργαζομένους, αλλά υπάρχει δημοψήφισμα και ο κρατικός λαός ε, απεφάνθη επισήμως και είπε ναι. Πώς θα γίνει, θα αρχίσουμε πάλι από την αρχή. Τρίτο και τελευταίο, η 1η Ιουλίου δεν είναι εφεύρημα δικό μας, αλλά υπάρχει σε μια συνθήκη που υπεγράφει από όλους τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Πώς θα κάνουμε δηλαδή, δεν είναι αυτά ε, πλασματικές ε, ημερομηνίες, είναι ημερομηνίες πραγματικές που υπάρχουν σε συνθήκη. Ευχαριστώ πολύ. Έχει δίκιο εις ό,τι αφορά την τυπική διαδικασία ο κ. Σπόσελτ Απεφάνθη θετικά με νομικά δεσμευτικό τρόπο το Κοινοβούλιο υπέρ της προσχώρησης της Κροατία. Οπότε εμείς έχουμε τελειώσει. Ε, ούτε μπορούμε ούτε θέλουμε να καθυστερήσουμε. Παρόλα αυτά όμως ε, έχει νόημα να βοηθήσει και η Κροατία και να ε, λύσει τα θέματα αυτά τα 10 γιατί μπορεί να υπάρξει εκκρεμότητα στην ακύρωση λόγω της καθυστέρησης εκεί. Και η Σλοβενία επίσης, γιατί πολλές φορές μπορεί να υπάρξουν εμπόδια στον επόμενο που θα έρθει. Με την παλιά θεωρία του λεωφορείου που μπαίνει ο τελευταίος, δεν πάει παραπέρα και λέει γέμισε το λεωφορείο, κλείνουν οι πόρτες. Η απεσιόδοξη εκτίμηση του συναδέλφου Σέπφλιν ελπίζω να μην ε, γίνει πραγματικότητα. Αλλά όλες οι πλευρές πρέπει να συνδράμουν θετικά. Και οι Κροάτες φίλοι επίσης. Να πληρούν τις προϋποθέσεις. κύριε Αμπράν. Ε, γυρίζω σε αυτό το τελευταίο θέμα για τις διμερείς ε, διαφορές. Ε, Κροατία, Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Σερβία ε, υπάρχουν διμερεί προβλήματα που επιμένουν. Πρέπει να βρούμε μια συνεκτική λύση και να είμαστε σοβαροί σε σχέση με το πώς εκτιμούμε τις διαφορές. Αποτελούν ε, προσκόμματα για να μην μπλοκάρει ο ένας τον άλλον. Να υπάρχει συνοχή λοιπόν και να ε, ξέρουμε και εμείς τι θέση θα λάβουμε ως Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν να μπλοκάρει, αυτή την μια γενική θέση, δεν μπορεί να μπλοκάρει ο τελευταίος ε, προσχωρήσας τον επόμενο. Κύριος Κασίν, ευχαριστώ. Συμφωνώ, αλλά θέλω και να προσθέσω κάτι. Αυτό που συζητάμε για την Κροατία και τη Σλοβενία δεν είναι θέμα διμερές. Είναι θέμα πολυμερές. Είναι θέμα διαδοχής. Η Κροατία συμφώνησε. Και αν διαβάσετε τη συμφωνία που υπεγράφει για την προσχώρηση της Κροατίας, ε, συμπεριλαμβάνεται. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι οι συνθήκες πρέπει να τηρούνται, πάκτα σουν σερβάντα. Όταν, στο βαθμό που η Κροατία δεν τηρεί τα υπεσχημένα, θα δυσκολεύεται. Και πιστέψτε με ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που μπορεί να εμποδίσει την Κροατία να προσχωρήσει στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, και αυτή είναι η τωρινή κυβέρνηση. Ε, και οι δύο πλευρές πρέπει να βρουν ε, μια λύση. Δεν σημαίνει ότι ένα κράτος μέλος που έχει βέτο θα πρέπει να κινηθεί κάποιο, άλλος, κάποιο άλλο όπως θέλουμε. Θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία και δεν μπορεί το κράτος μέλος να εκμεταλλεύεται το βέτο που έχει. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει προθυμία και ετοιμότητα για λύση και από τις δύο πλευρές. Αυτό ισχύει γενικά για τέτοιου είδους διαφορές. Ο κύριος Σαγκουράκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να πω στον κύριο Πόσελ. Βεβαίω έχει δίκιο, το ξέρω αυτό. Αλλά με μια μικρή διαφορά. Η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι εκείνη που ψήφισε υπέρ της προσχώρησης. Ξέρω πολύ καλά το αποτέλεσμα του κροατικού δημοψηφίσματος, γιατί πήγα στη χώρα και μίλησα και με τον κόσμο και με τις πολιτικές δυνάμεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όταν ε, υποβληθεί η έκθεση για τη χώρα αυτή ότι δεν μπορούμε να εκφράσουμε τη γνώμη μας. Αυτό έκανα. Είμαι ευγνώμων στον εισηγητή για την έκθεσή του, γιατί κατά τη γνώμη μου με ενισχύει στην πεποίθησή μου ότι η προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν εξυπηρετεί τη μεγάλη πλειοψηφία των Κροατών. Τίποτε περισσότερο. Ευχαριστώ. Συνάδελφε, κανείς δεν σας εμποδίζει να εκφράσετε την όποια γνώμη σας. Ο κύριος ε, Λάγκεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα με αυτή την ευκαιρία να ενημερώσω τι κάνει η Κομισιόν τώρα σε σχέση με την παρακολούθηση της χώρας αυτής ε, της Κροατίας. Ε, το σχέδιό μας είναι να ε, δώσουμε την νεαρινή έκθεση στις 21 Μαρτίου όπου θα επιμείνουμε στα τρία κυρίως κεφάλαια, το 8 για τον ανταγωνισμό, 23 και 24 που καλύπτουν όλο το θέμα του κράτους δικαίου Επίσης ζητήσαμε πληροφορίες από την Κροατία να μας πούν ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Τα στοιχεία αυτά τα αναλύουμε τώρα και έγινε και συνεδρίαση μεταξύ του Επιτρόπου Φίλε και της Υπουργού Εξωτερικών Πούσιτς την περασμένη εβδομάδα και από την κροατική πλευρά ενημερώθηκε ο Επίτροπος για τις τελευταίες εξελίξεις. Γενικά η αντίδραση του κυρίου Φίλε ήταν να εκφράσει την ικανοποίησή του με τις πρόοδους που επιτελούνται στην Κροατία και τους ενθαρρύνει να κάνουν και την υπόλοιπη δουλειά μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης. Ε, κάνοντας μια προσωρινή εκτίμηση μπορούμε να πούμε ότι τρία από τα δέκα σημεία δημιουργούν δυσκολίες και είναι δύσκολο να τα έχουν προλάβει μέχρι την ιαρινή έκθεση. Το ένα ε, είναι η ιδιωτικοποίηση των ναυπηγείων. Ε, χθες, έγινε συζήτηση μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και του, της Κροατίας και του Επιτρόπου Αλμούνια και από ό,τι κατάλαβα ε, μια συμφωνία ότι η Ευρωπαϊκή, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει τώρα νέα ε, απόφαση. όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και στον Board Split που θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά, θα υπάρξει γενικότερη αναφορά στα ναυπηγεία θετική στην έκθεση της Άνοιξης. Το δεύτερο θέμα που μάλλον δεν θα το καταφέρουν να το τελειώσουν είναι αυτό το, αυτή η συνοριακή διάβαση του διαδρόμου του νέου. Έχουν αρχίσει οι εργασίες ε, πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά δεν θα έχουν ολοκληρωθεί. Δεν γίνεται μέχρι το Μάρτιο. Εμείς υποθέτουμε και τώρα παίρνουμε πληροφορίες από την Κροατία που δείχνουν ότι θα προχωρήσουν ε, οι εργασίες σε αυτό το τομέα, ούτως ώστε να είναι έτοιμοι όταν θα είναι η Κροατία έτοιμη να προσχωρήσει. Η μεταφράση τέλος, η κροατική γλώσσα θα είναι μια επίσημη γλώσσα και πρέπει όλο το κεκτημένο να μεταφραστεί στα κροατικά από τους Κροάτες. Είναι μεγάλη δουλειά αυτή, μακράς πνοής. Κατά τη διάρκεια αυτή την εβδομάδα θα γίνουν συνεδριάσεις με τα αρμόδια μεταφραστικά γραφεία των Κροατών, ούτω ώστε να δούμε πού είναι τα πράγματα. Από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι έτοιμα όλα μέχρι την έκθεση του Μαρτίου, αλλά θα προσπαθήσουμε να μάθουμε μήπως προλαβαίνουν να τελειώσουν μέχρι την 1η Ιουλίου με ενημερώνουν ότι προέκυψε ένα θέμα ακόμη σχετικά με τη διαφορά ή το ζήτημα Μαυροβουνίου-Κροατίας, γιατί υπάρχει θέμα συνόρων και εκεί, στο ε, Χερσόνησο Πρεφλάκα. Εκεί, από ό,τι με διαβεβαιώνουν ε, σε διμερές επίπεδο, γίνονται συνομιλίες μεταξύ Κροατίας και Μαυροβουνίου για την εξέβραση λύσης το θέμα ετέθη χθε και από τον πρόεδρο Μπαρόζο όταν, όταν συνάντησε τον πρωθυπουργό Τζουκάνοβιτς ε, του Μαυρονίου και ε, υπάρχουν ενθαρρύνσεις στο ώστε σύντομα να ξεβρεθεί λύση και στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ο εισηγητής κ. Ρούτσεκ για Έχετε το λόγο για τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα επικοδομητικά σας σχόλια και για τις ε, κριτικές σας ίσως ε, να πρέπει να ανατρέξω ένα σημείο της παρατηρήσης. Κύριε Πόσελτ, ε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας πως είναι ε, η δουλειά και η επιτυχία όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά όλων των πολιτικών δυνάμεων. Αν μια χώρα, άσχετα με το αν είναι Κροατία, Μαυροβούνιο, οποιαδήποτε χώρα θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία όλων των βασικών πολιτικών δυνάμεων και αυτό ακριβώς συμβαίνει στην Κροατία. Όπως ήδη ανέφερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω δε και να συγχαρώ τους παρατηρητές μας από όλες τις πολιτικές ομάδες για την δουλειά τους, την συμβολή τους στις εργασίες μας, όχι μόνο στην ΑΦΕΤ, την Επιτροπή δηλαδή Εξωτερικών, αλλά και στο σύνολο του Κοινοβουλίου. Ε, κύριε Κατσίν, επικύρωση, θα το αναφέρω στο τέλος. Κυρία Μπραντνερ, κράτος δικαίου. Διαφθορά, δημόσια δίκηση, εγκλήματα πολέμου. Αυτά είναι σημεία που εστιάζω την προσοχή, όπως ήδη ανέφερα, ναι, ορισμένα πράγματα πρέπει να γίνουν πριν την ένταξη. Αλλά είναι μια ε, διαδικασία υπό εξέλιξη. Όπως και το παράδειγμα όλων των υπόλοιπων ε, ε, νέων κατρομελών συμπεριλαμβανωμένες και στις χώρες μου. αναφέρεται πως η Κροατία είναι έτοιμη ε, Ακριβώς σε αυτό το θέμα και εγώ εστίασα την προσοχή μου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στην Κροατία. Το τόνισα για, παίρνοντας σαν παράδειγμα τη χώρα μου, την Τσεχία που είναι μέλος εδώ και ένα χρόνια και λόγω της διαφθοράς δεν μπορεί απόλυτα να επωφεληθεί, να χρησιμοποιήσει τα χρήματα και να αυξήσει το οικονομικό της δυναμικό. Οι Κροάτες φίλοι λοιπόν το γνωρίζουν, εργάζονται από αυτού και διαρκώς βελτιώνουν την κατάσταση. Επίσης ξέρουν ότι δεν πρόκειται να, να τελειώσει αυτή η δουλειά 1η Ιουλίου. Είναι μια διαρκής μόνιμη διαδικασία. Έπειτα ε, το έχω αναφέρει πολλές φορές και εσείς το επαναλάβατε, ότι χρειάζεται δηλαδή περισσότερη δουλειά, περισσότερη παρακολούθηση από το Κοινοβούλιο της χώρας και το ίδιο ισχύει για την κοινωνία των πολιτών. Να συμμετέχει δηλαδή η κοινωνία των πολιτών στην καθημερινή δουλειά του Κοινοβουλίου. Κύριε Τάνοκ, συνοριακή διαμάχη ανάμεσα στην Κροατία και στο Μαυροβούνιο. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε σχέση με τα όσα είπε ο, συνάδελφος, ο κύριος της συνάδελφος της Επιτροπής. Έχω λάβει ε, διαβεβαιώσεις από τα διάφορα μέλη της, της κυβέρνησης της Κροατίας, αλλά συμφωνώ ότι πρέπει να παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή, ώστε να μην έχουμε εκπλήξεις ούτε τώρα ούτε και αργότερα διότι είναι προς το συμφέρον της Κροατίας, προς το συμφέρον του Μαυροβουνίου και του συνόλου της διαδικασίας διεύρυνσης. Όσον αφορά αυτά τα εναπομείνοντα διμερεί θέματα, όχι ανάμεσα στην Κροατία και το Μαυροβούνιο μόνο, αλλά στα Βαλκάνια γενικότερα, θα πρέπει να λύνονται όσο γίνεται πιο σύντομα. Και από ό,τι καταλαβαίνω, είναι και τμήμα της νέας στρατηγικής της Κομισιόν και του Επιτρόπου για ολόκληρη την περιοχή. Κύριε Κούκαν, η ε, μεταρρυθμίσει του δικαστικού σώματος, οι μεταρρυθμίσει των κρατικών προμηθειών και αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα, το τονίζω. Κύριε Γκουράκη, δεν συμφωνώ μαζί σας όσον αφορά το σημείο 13 της έκθεσης, διότι τι λέει. Ενθαρρύνει την Κροατία να προβεί σε διαρθρωτικές αλλαγές για να κινητοποιήσει την οικονομική αγορά και να αποκαταστήσει την αγορά εργασίας. Μα πώς αλλιώς να κινητοποιηθεί η ανάπτυξη χωρίς μεταρρυθμίσεις. Έχουμε θετικά και αρνητικά παραδείγματα από πολλές χώρες που έχουν ε, κάνει μεταρρυθμίσεις είτε από την από αριστερή κυβέρνηση είτε από δεξιά. Χωρίς διαρθωτικές αλλαγές δεν γίνεται οικονομική ανάπτυξη και χωρίς οικονομική ανάπτυξη δεν υπάρχει αύξηση στην απασχόληση. Πραγματικά δεν... Πιστεύω πως κάτι τέτοιο θα οδηγήσει στην ανεργία. Όπως είπα, έχουμε πολλά καλά παραδείγματα. Δείτε την Αυστρία, δείτε τη Γερμανία, δείτε κάποια από τα νέα κρατημέλη ή από τη Σλοβακία είτε από τη Σλοβενία. Οι χώρες κινούνται, έχουν οικονομική ανάπτυξη ακόμα και σε μια φάση που πολλά κρατημέλη συμπεριλαμβανομένου του δικού σας ε, βρίσκονται σε κρίση. Εγώ θα πρότεινα να δείτε αυτές τις θετικές, τα θετικά παραδείγματα και προσπαθήστε να τα εφαρμόσετε και στην χώρα σας. Τώρα, 18. Σημείο 18 ανεφέρθη ότι ο Πρωθυπουργό Μιλάνοβιτς συναντήθηκε με τον Σέρβο Πρωθυπουργό στο και Ακριβώς αυτά τα θέματα συζήτησαν την ε, θέση των κρατικής μειονότητας στην Κροατία, την δίωξη των ε, εγκλημάτων πολέμου, την επιστροφή των προσφύγων, συνοριακά θέματα και ούτω καθεξής. Οπότε, ναι, νομίζω πως και οι δύο πλευρές γνωρίζουν το πρόβλημα και εργάζονται. Και αναφέρατε και το σημείο 21. 21 όπου έχουμε κάποια διμερεί θέματα όπως ήδη ανέφερα ναι, θα πρέπει να εστιάσουμε στην επίλυση των διμερών ζητημάτων και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά επηρεάζουν ολόκληρη την περιοχή αυτή. Αναφέρατε την ομάδα σας και ότι εσείς ε, είστε κατά της προσχώρησης της κουρατίας. Δεν το καταλαβαίνω εγώ πιστεύω πως είναι προς το συμφέρον ολόκληρη της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της χώρας σας, να επικρατεί σταθερότητα στην Ευρώπη. και η προσχώρηση της Κροατίας σίγουρα θα συμβάλλει στην αύξηση της σταθερότητας σε αυτή την ιδιαίτερα σταθή περιοχή της Ευρώπης στα Βαλκάνια και θα είναι θετικός ο αντίκτυπος για τις χώρες και για τη δική σας χώρα. να μιλήσω για τον κύριο Σέφλιν και για το θέμα της υπολοιπόμενης επικύρωσης. Δεν συμφωνώ μαζί σας με το σχέδιο Β αν πληρωθούν οι προϋποθέσεις, οι όροι. Το είπα και ο κύριος Πόσελ και τον έφερε και ο πρόεδρος μας ότι υπάρχουν κάποια νομικά δεσμευτικά θέματα να τονίσω φιλικά ότι η Ουγγαρία και οι Ούγγροι είναι γνωστοί ως πολύ απεσιόδοξοι τύποι. Πολύ δύσκολο να τα αλλάξουμε αυτό. Το ξέρω, αλλά ας είμαστε θετικοί, ας είμαστε αισιόδοξοι, ας δουλέψουμε όλοι μαζί ε, ώστε την 1η Ιουλίου η Κροατία να γίνει μέλος της Ένωσης. Δηλαδή, Κανένας δεν δουλεύει για σχέδιο Β. Κανένας δεν σκέφτεται το σχέδιο Β. Η δέσμευσή μας ε, και όλων των φίλων της Κροατίας είναι να είναι μέλη την 1η Ιουλίου. Και πάλι πρέπει να τονίσω πως είναι προς το ζωτικό συμφέρον της Ουγγαρίας, της χώρας σας, να γίνει κάτι τέτοιο. Και της χώρας σας μάλλον. Now still, still the last about... Λοιπόν, τελευταία λέξη μου για την επικύρωση και τη Σλοβενία. Είναι λογικό η Σλοβενία, μια φιλική χώρα που είναι γείτονα τη Κροατία. να κινηθεί σε αυτή τη θέση της τελευταίας. Γιατί Ακριβώ για αυτό το πράγμα μιλάμε, ότι οι χώρε τη πρώην Ιουγκοσλαβία να είναι στην πρωτοπορία, να είναι οι πρωτεργάτες της περαιτέρω διεύρυνσης. Και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ακόμα πολλά εκκρεμισδήματα, δήματα, διμερεί, αλλά και πάλι ας δούμε το θέμα από θετική σκοπιά. Είναι ζωτικό συμφέρον της Σλοβενίας η Κροατία να είναι μέλος. Αν λάβετε υπόψη τι θα συμβεί στη διαδικασία διεύρυνσης Κροατίας-Σλοβανία, αν μπλοκαριστεί αυτή η κατάσταση, κανένα δεν θα βγει κερδισμένος. Ούτε η Κροατία, ούτε η Σλοβενία, ούτε και η Ευρώπη. Ας δουλέψουμε λοιπόν θετικά προς την επίλυση του προβλήματος. Χτες έγινε συνάντηση των δύο εμπειρογνωμών, δεν ξέρουμε αν θα βρεθεί λύση. Εάν βρεθεί, τόσο το καλύτερο. Εάν όχι, εξαρτάται και από τις δύο κυβερνήσεις να βρουν λύση όσο γίνεται πιο σύντομα. Γιατί όπως είπα, δεν είναι προς το συμφέρον της Σλοβενίας ούτε προς το συμφέρον της Κροατίας. Ας δουλέψουμε προς, προς το στόχο της πρώτης Ιουλίου. Γιατί αν δεν γίνει αυτό θα είναι μακρόπνες οι επιπτώσεις και για τη Σλοβενία και για ολόκληρη την περιοχή. Τελευταία μου λέξη. Μην ξεχνάτε τις ε, διαφορές που είχε η Σλοβενία με την Ιταλία. Αν η Ιταλία είχε συμπεριφερθεί με, με, τέτοιο τρόπο, δεν θα μιλούσαμε τώρα για την ε, Κροατία, αλλά για τη Σλοβενία. Ας το έχουμε αυτό υπόψη, λοιπόν. Κύριος Κατσίν, ένα σύντομο σχόλιο, παρακαλώ. Μάλιστα. Προσωπικά μου, μίλησε ο προσωπικός μου φίλος και συνάδελφος ότι η Σλοβενία θα έπρεπε να είναι ανάμεσα στους πρώτους που θα επικυρώσουν τη συμφωνία προσχώρησης με την Κροατία. Αλλά δυστυχώς έχει γίνει κάτι εντωμεταξύ και το μπλοκάρισμα είναι συνέπεια αυτού και χρειάζεται να απεμπλακεί η κατάσταση. Εκτιμώ και καλωσορίζω την πρόσφατη πρωτοβουλία και δήλωση του Πρωθυπουργού Κούσιτς, ο οποίος ζητά να βρεθεί μια διέξοδος. Και νομίζω πως μπορεί να βρεθεί η διέξοδο. Σας είπα ποιος είναι ο τρόπος να βγούμε από το πρόβλημα. Και από τη στιγμή που θα υπάρχουν αυτοί οι όροι, θα πληρούνται οι όροι, η Σλοβενία θα κάνει τη δουλειά της. Να υπογραμμίσω και πάλι πως είναι στρατηγικό συμφέρον της Σλοβενίας να έχει άμεσο γείτονα. Θέλουμε την Κροατία, όχι μόνο απλά στην Ένωση, αλλά στο Σέγγεν και να πάψουν οι έλεγχοι του Σέγγεν ε, όσο γίνεται πιο σύντομα. Είμαστε στα δικά μας σύνορα. Εγώ λοιπόν σας παρακαλώ να μας πείτε πώς μπορούμε να απεμπλέξουμε αυτήν την κατάσταση ώστε να γίνει όσο αυτό όσο γίνεται πιο γρήγορα. Παρά την κρίση στη Σλοβενία πιστεύω πως όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε και ακόμα και αν χάσουμε την κυβέρνηση, το κοινοβούλιο δεν θα διαλυθεί και θα κάνω τη δουλειά τους εγκαίρως. Ας κάνουμε λοιπόν κάθε πλευρά το τμήμα της εργασίας που της αναλογεί. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Να σας θυμίσω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 24 Ιανουαρίου, το μεσημέρι στις 12. ψήφισμα, πρόταση ψηφίσματο για την έκθεση προόδου 2012 για την πρώην Ιγκοσλαβική Δημοκρατία της ε, Μακεδονίας. Ο εισηγητή είναι ο κύριος Ρίτσαρντ Χόουιτ. Έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Πρόκειται για την πρώτη εξέταση του σχεδίου Έκθεση για την πρόοδο της πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατίας τη Μακεδονία και είναι ένα από τα νέα ψηφίσματα που λάβαμε. Το Δεκέμβριο, που γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να καλέσει την Κομισιόν να παρουσιάσει την άνοιξη του 2013 μια έκθεση για την εφαρμογή των την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των βημάτων που έχουν σημειωθεί για τη βελτίωση των ε, σχέσεων ίαση. Ε, από αυτέ τι βάσει, το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να ξεκινήσει ενταξιακέ διαπραγματεύσει με τη χώρα αυτή. Το σχέδιο ψηφίσματο εξετάζει έναν αριθμό προκλήσεων κλειδιών στη διαδικασία προσχώρηση αυτή τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών κριτηρίων της κοινωνίας των πολιτών, οικονομικά ζητήματα, αλλά και βήματα ως ώστε να βελτιωθούν οι σχέσεις γετνίασης αλλά και η περιφερειακή συνεργασία. Κύριε Χάουιτ, που είστε εισηγητής, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλημέρα σας και θα ήθελα να ξεκινήσω ε, σχολιάζοντας σύντομα δύο επίκαιρα θέματα, διότι ο στόχος της έκθεσής μας δεν είναι να κοιτάμε προς τα πίσω, αλλά προς τα εμπρός. Και γι' αυτό η δουλειά μου ήταν να προσπαθήσω να ε, τονίσω και να φωτίσω το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας. Όπως θα γνωρίζετε, συνάδελφοι, υπήρξε μια σύγκρουση ανάμεσα στα μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα της χώρας πριν τα Χριστούγεννα, όταν συμφωνήθηκε ο προπολογισμό στο Κοινοβούλιο με αντιφατικό τρόπο γιατί το κόμμα της αντιπολίτευσης έφυγε, αποχώρησε από το Κοινοβούλιο και έκτοτε κάνει διαμαρτυρίες στους δρόμους έχουν κινητοποιηθεί 70 με 100.000 άνθρωποι στους δρόμους των Σκοπίων. Τελικά φαίνεται να... ότι θα ξαναγίνει συζήτηση στο Μάρτιο. Προσπάθησα να είμαι πολύ προσεκτικός και να μην ε, ε, μπορεί να κατηγορηθεί το Κοινοβούλιο για παρέμβαση στην εθνική πολιτική της χώρας. Αλλά πιστεύω πως είναι σημαντικό να πούμε σε όλα τα πολιτικά κόμματα της χώρας ότι αν θέλουμε να υπάρξει πρόοδος πράγμα που εγώ σίγουρα επιθυμώ για τη χώρα αυτή, σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινοβούλιο ε, ε, δυνατό, στεναρό, που όλα τα χώρα, όλα τα κόμματα συμμετέχουν εκεί και όπου υπάρχει σεβασμός για όλα τα πολιτικά κόμματα, τα κυβερνητικά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και φυσικά είναι σημαντικό να υπάρχει πολιτικός διάλογος, πολιτική πειθαρχία, αλλά φυσικά στο πνεύμα ενός ε, διαλόγου ανάμεσα στα κόμματα. Και σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα απλά να σας αναφέρω, συνάδελφοι, γιατί μπορεί να μην το γνωρίζετε, πως εχθές ο Πρωθυπουργό της χώρας εξέδωσε μια πρόσκληση προς την αντιπολίτευση, ώστε να συνεχίνουν ε, ε, πρόσωπο με πρόσωπο συνομιλίες για πρώτη φορά μετά από, αυτές τις, από αυτά τα γεγονότα. Και σήμερα γίνεται αυτή η συνάντηση στα Σκόπια. Η αντιπολίτευση δέχτηκε την πρόσκληση και ήδη αυτό δείχνει ένα πνεύμα προόδου θέλουν η χώρα τους να προχωρήσει προς τις ε, διώξεις και τις ε, φιλοδοξίες για ένταξη στην Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Αυτά λοιπόν αυτά είχα να σας πω αρχικά και να πω σε αυτούς που θα ήθελα να χρησιμοποιήσουν αυτή την πολιτική κρίση ως ε, περαιτέρω λαβή για αντιρρήσεις ή για να μπλοκάρουν την πρόοδο της χώρας Ελπίζω λοιπόν ότι θα δούμε πως η συγκεκριμένη κρίση έχει ξεπεραστεί και ότι τελικά θα φανεί η δύναμη της δημοκρατίας και των θεσμών στη χώρα. Έχουν υποχρέωση ε, να το καταφέρουν αυτό, αλλά και εμείς το ίδιο. Η δεύτερη μου παρατήρηση έχει να κάνει με τον Επίτροπο Στέφαν Φίλου που ήδη έχει πει δημόσια ε, πήρε μια πολύ τολμηρή θέση όταν ήρθε εδώ το Θευθυνόπορο για να μας παρουσιάσει την έκθεση πρόοδου και είπε ότι εκείνο ω Επίτροπο θα αλλάξει τη θέση τη Κομισιόν και ότι θα προχωρήσει, προωθήσει μάλλον την ιδέα του ζητήματο του ονόματο και την επίλυση αυτού που δεν, όχι πριν από την ένταξη της χώρας, αλλά στα πρώτα σε φάσεις ε, των διαπραγματεύσεων. Φυσικά οι Έλληνες συνάδελφοι δυσκολεύτηκαν όταν το άκουσαν αυτό, αλλά και οι υπόλοιποι Έλληνες. Αλλά δεν ήταν ε, μια προσπάθεια να παραβιάσει το status quo. Δεν ε, έρει την υποχρέωση όσων ε, βρίσκονται στη χώρα ώστε ε, να ξεκινήσουν οι πραγματεύσεις ε, καλή την πίστη ώστε να βρεθεί μια αποδεκτή λύση αλλά προσέφερε την ε, προοπτική για αλλαγή και εγώ το στηρίζω αυτό. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που το, Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου δεν παρατήρησε απλά τη θέση, δεν κράτησε την ίδια θέση που είχε πριν τρία χρο... εδώ και τρία χρόνια, αλλά ζήτησε μια ακόμα έκθεση μέχρι τον Ιούνιο φέτος, όπως είπατε Πρόεδρε, ώστε να ληφθεί απόφαση στο πρώτο ήμιση του έτους. Και εγώ καλωσορίζω το βήμα αυτό γιατί πιστεύω πως δίνει όντως μια νέα ευκαιρία και είναι μια ευκαιρία μάλιστα που αν όλοι μας την εκμεταλλευτούμε, μάλλον που αν δεν την εκμεταλλευτούμε τώρα μπορεί να μην την έχουμε και πολύ σύντομα ξανά. Αυτά λοιπόν και τώρα θα σας πω δύο λόγια για το σχέδιο εκθεσής μου. Εγώ στην έκθεσή μου εκτιμώ τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου και λέω ότι μπορεί η έναρξη των διαπραγματεύσεων να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο και να αλλάξουν την κατάσταση. Όσοι λένε πως δεν ήρθε ακόμα ο καιρός, ε, θα πρέπει να καταλάβουν πως υπάρχει σχέση ανάμεσα στην στη γνήσια προοπτική προς ε, ενταξιακή διαπραγμάτευση και την κατάλληλη στιγμή για τις μεταρρυθμίσεις. Εγώ πιστεύω πως τα κριτήρια πληρούνται επαρκώς και αν θέλουμε πραγματικά να υπάρξει επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στη χώρα θα ήταν σωστό να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις ώστε να μπορέσει να συμβεί αυτό. Επίσης σημειώνω την ε, λειτουργία του διαλόγου και ήταν επιτυχής. Το 75% των ε, τομέων πολιτικής που έχουν εντοπιστεί στο τριμερή διάλογο από την Κομισιόν έχουν ε, σημειώσει πρόοδο. Η τρίτη μου παρτήρηση είναι ότι ζητώ από την Κομισιόν όταν παρουσιάζει τις εκθέσεις να μην αναλύει απλά τη χώρα και την πρόοδο της, αλλά να αναλύει και το κόστος της μη διεύρυνσης, της μη πρόοδου δηλαδή. Αυτό μπορεί να αληθεύει και για άλλες χώρες στην Ευρώπη στην περιοχή. Αλλά σίγουρα αληθεύει για αυτήν εδώ. Και ένα τέταρτο χειρισμό αφορά την Ιρλανδική Προεδρία, γιατί έχω, έχω υποστηρίξει τον Επίτροπο Φίλου, αλλά η Ιρλανδική Προεδρία είπε, δήλωσε ότι θέλει να υπάρξει πρόοδος στην χώρα και εγώ τους κάνω έκκληση ώστε όντως να ε, υπάρξει αυτή η πρόοδος. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Στην, στην παρουσίασή μου υπάρχουν κοινά στοιχεία από την έκθεσή μου πέρυσι. Για το θέμα του ονόματος, μια ωραία πρόταση από τους πράσινους πριν από τρία χρόνια, αλλά που το έχουμε ξανασυζητήσει έκτοτε θα έπρεπε να ασκήσετε μια κάποια πίεση από την Ένωση για να λύνονται τα διμερεί θέματα και στην παράγραφο 1 λέω πως θα πρέπει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις άνευ Αυτή είναι η θέση του Κοινοβουλίου, όχι του Συμβουλίου και να το επαναλάβω ότι φέτος 600 βουλευτές το υπερψήφισαν αυτό και αυτό τονίζει και ασκεί πίεση και καθώς και δίνει ένα μήνυμα. και πάλι αυτοί που θέλουν να κεφαλοποιήσουν πολιτικά την κρίση ε, να σας πω ότι ήταν τεράστια η κρίση ανάμεσα στα δύο κυβερνητικά κόμματα τον Αύγουστο και κάποιες εβδομάδες μετά. Ε, δεν λέω ότι λύθηκε, αλλά έχει ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι μια καλή, ένα καλό σημάδι για την στεναρότητα της δημοκρατίας στη χώρα έχει υπάρξει μείωση και των δικαστικών υποθέσεων καθώς και περισσότερη ελευθερία τύπου. Ε, ε, αλλά όχι επαρκής. Αυτό θα πρέπει να μας ανησυχεί. Μιλάω για τα θέματα των διακρίσεων, για την οικονομική πρόοδο και τις μόνιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, που όλοι αντιμετωπίζουμε δηλαδή από την ευρωπαϊκή και οικονομική παγκόσμια κρίση που είναι κατά τη γνώμη μου το μεγαλύτερο κίνητρο για τη χώρα αυτή να μπει στην Ένωση ε, φέτος τώρα Προσπαθώ να εξετάσω κάποια συγκεκριμένα τμήματα της έκθεσης και να μην δώσω γενική εικόνα ε, μόνο και να πιέσω δηλαδή για ορισμένα θέματα. Ως εισηγητής έχω επισκεφτεί τη χώρα πολλές φορές και θα σας πω ότι κάθε φορά είχα ένα θέμα. Ε, ερχόμουν σε επαφή από τον με τον κόσμο της πολιτικής αλλά και με την κοινωνία των πολιτών θέματα όπως ε, η διαφθορά, η αποκέντρωση, η παιδεία συμπεριλαμβανομένης ε, της ένταξης ε, των παιδιών με ειδικές ανάγκες και της πολυεθνικής παιδείας και πρότεινα στην Επιτροπή, στο Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν να δοθούν περισσότερα χρήματα στην και περιφερειακή ε, κυβέρνηση και να συγχαρώ μάλιστα τη UNDP που έχει στηρίξει πολύ την περιφερειακή και τοπική κυβέρνηση και, θα, και κάναμε και ένα, μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζας με εκπροσώπους, 30-40 μάλλον εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών πριν συντάξω την εκθεσή μου και εκεί υπήρξαν διάφορες προτάσεις που σας τις υποβάλλω για την ενίσχυση της, ανεξα... της ανεξαρτησίας και του πλουραλισμού οι ίδιες οι οργανώσεις της κοινωνίας ε, θα πρέπει να προστατέψουν την ανεξαρτησία τους. Είναι πολύ σημαντικό σε μια πολύ πολιτικοποιημένη χώρα και περιβάλλον. Ζητούν οι ομάδες εργασίας της κυβέρνησης να έχουν επαφή με την κοινωνία των πολιτών, ζητούν τις διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών και Ε, μέσα ώστε να μπορέσουν οι οργανώσεις της κοινωνίας να εκμεταλλευτούν τα χρήματα που δίνονται και το 15 μάλιστα των χρημάτων που δίνονται στην χώρα να δίνονται στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Να υπάρξει δηλαδή συνεργασία και με άλλες ε, και ΜΚΟ ε, στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία κτλ. Τέλος, ε, Πρόεδρε, θα υποβάλω στην Επιτροπή κάτι που έκανα και πέρσι και που είχε επιτυχία, να γίνει μια διαδικαστική τροπολογία, όταν ξεκινήσει η ψηφοφορία, δηλαδή να μην παίξουμε παιχνίδια σε αυτήν την Επιτροπή όπου κάποιοι θα λένε ότι θα, να βάζουμε όσο γίνεται περισσότερο που γουδουμό όσο γίνεται περισσότερο, ενώ οι άλλοι να λένε όχι θα βάλουμε Μακεδονία όσο γίνεται περισσότερο και τελικά όλοι να ε, κνευρίζονται με τα αποτελέσματα. Αυτό δεν αντικατοπτρίζει το Κοινοβούλιο και δεν θα βοηθήσει την Ελλάδα ούτε και την ε, που δούμε να υπογράψουν λύση. Λοιπόν, προτείνω λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε το όνομα που είναι το όνομα που γίνεται σεβαστό σύμφωνα με τη συμφωνία του ΟΗΕ, δηλαδή πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, χρησιμοποιείται, χρησιμοποιείται μία στον τίτλο και να χρησιμοποιούμε την λέξη Μακεδόνα, μακεδονική μόνο μία φορά στο κείμενο, γιατί αυτό σημαίνει ότι ζητάμε από την Κομισιόν, όπως και ο ΙΕ, να χρησιμοποιείται αυτή η λέξη, ώστε να αντικατοπτρίζονται όλες οι γλώσσες και οι εθνικές μειονότητες της χώρας με αυτή τη λέξη. Εχτε, πέρυσι τα πήγαμε καλά και ζητώ να γίνει το ίδιο και φέτος. Για τους βούλγαρους φίλους βλέπω τον κύριο Κυρίλο Φεδό και τον κύριο Κόβατσοφ. είχατε τι συζητήσεις μαζί σας πέρυσι και για τη διάρκεια του περασμένου έτους και σιώπησα εδώ για διάφορα θέματα. Ξέρω πώς είναι σημαντικά για εσάς γιατί την κοινή, κοινό εορτασμό ιστορικών γεγονότων, την ταυτότητα, τον, την βουλγαρική μειονότητα στη χώρα. Δεν υποτιμώ τη σημασία αυτών των θεμάτων. Ξέρω πώς θα υποβάλλετε τροπολογίες και θα υποβάλλω και εγώ τις δικές μου. Θα κάτσουμε μαζί λοιπόν και θα βρούμε μια συμβιβαστική δίκαιη ε, όπως κάναμε και πέρσι. Αλλά πιστεύω Και να πω και στην κυρία Κοπά και στους Έλληνες συνάδελφους που είναι εδώ ότι το Ελληνικό Υπουργείο ανταποκρίθηκε στην τριμερή συνάντηση που πρότεινε ο Επίτροπος Φίλε ε, αυτή την εβδομάδα. Θα υπάρξει συνάντηση για το θέμα του ονόματος, όχι για να το επιλύσουμε, όχι παράλληλα με τον ΟΙΑ, αλλά για να στηριχτεί ε, η λύση και το ότι το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δέχτηκε αυτή την πρόσκληση επί τη βάση του ότι η Ελλάδα πιστεύει πως μπορεί να υπάρξει ένα αποτέλεσμα. Και το λέω λοιπόν στους Έλληνες φίλους και την κυρία Κόπα ότι εγώ καλωσορίζω αυτή τη θέση της Ελλάδας και πρέπει όλοι να ελπίζουμε πως αυτή η τριμερή συνάντηση θα οδηγήσει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα προς την επίλυση της διαφοράς. Πρόεδρε, μόλις είχαμε μια συζήτηση για την Κροατία και μάλιστα συμμερίζομαι την άποψη της πλειοψηφίας ότι η 1η Ιουλίου είναι μια ημερομηνία που δεν μπορεί να μετακινηθεί και είπε ε, ο εισηγητής Ρούτσικ ότι δεν υπάρχει πλάνο σχέδιο Β και το ίδιο θέλω να σας ζητήσω και για αυτήν εδώ τη χώρα, την ε, Φύρομ. Δεν υπάρχει σχέδιο Β έχει μείνει σε ένα λίμπο, σε μια αοριστία. Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία μας τον Ιούνιο να το διευκολύνουμε αυτό προς το συμφέρον της χώρας, του λαού. για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να υπάρξει μια αλλαγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χόβιτ. Πρώτος στον κατάλογο μιλητών είναι ο κύριος Κόκαν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την έκθεση και συγχαρητήρια στον εισηγητή για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε και αφοσιώθηκε σε αυτό το θέμα για τη Μακεδονία. Η έκθεση αναφέρει όλα τα σημαντικά σημεία που έχουν να κάνουν με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ατζέντα για τη Μακεδονία. Η χώρα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά πρέπει να πληρώσει το τίμημα για ένα άλλο θέμα που παραμένει με τους γειτονές της. Αυτή είναι μια κατάσταση δίχως ε, προηγούμενο που κρατάει τόσα πολλά χρόνια και έχει βάλει τη χώρα και την περιοχή κατά κάποιο τρόπο ολόκληρη σε μια κατάσταση που πάει πίσω η διαδικασία ολοκλήρωση στην περιοχή και δεν ε, βοηθάει και την γενικότερη κατάσταση εκεί. Και παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει πολλά τελευταία για να ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση, παραμένει. Η έκθεση κάνει έκκληση στην Επιτροπή και το Συμβούλιο να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις όσο γίνεται πιο γρήγορα. Το στηρίζω αυτό, όπως επίσης και την πρωτοβουλία του Επιτρόπου Φίλε και των συνεργατών του και την ανορθόδοξη προσέγγιση του όσον αφορά τη διαδικασία ολοκλήρωση. Ο διάλογος ε, πάντως και οι συνομιλίες, ο ενταξιακός διάλογος έχουν αποφέρει αποτελέσματα, όπως όμως λέει και η έκθεση, δεν αντικαθιστά τις συνομιλίες για ένταξη. Πρέπει όλα αυτά να μπουν στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για να στηριχθεί και η δημοκρατική μετάβαση και οι μεταρρυθμίσεις στη χώρα αυτή. Η ατζέντα για τη διεύρυνση ε, περιλαμβάνει πολλά εργαλεία για να στηρίξουμε τις δημοκρατικές εξελίξεις στη χώρα και νομίζω ότι θα έπρεπε ήδη να είχαν χρησιμοποιηθεί εκεί. Στηρίζω επίσης την ιδέα του μηχανισμού διαιτησίας, ο οποίος ε, έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες εκθέσεις και ο οποίος ε, θα επιλύσει, ελπίζουμε, προβλήματα που αντιμετωπίζει με διμερεί θέματα η Μακεδονία σήμερα. Το θέμα του προπολογισμού του 2013 και επιπτώσεις στο Κοινοβούλιο και γενικότερα έχουν οδηγήσει τη χώρα σε δύσκολες καταστάσεις, σε δύσκολα νερά. Όπως δείχνουν τα πράγματα, όσο μπλοκάρεται η θεσμική συνεργασία μεταξύ της αντιπολίτευσης και του συνασπισμού, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πάει πίσω τη χώρα. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι πρέπει να στηρίξουμε όλες τις πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ως στόχο να ε, προχωρήσει ο διορθωμένος διάλογος για να προχωρήσει δημοκρατικά η χώρα. Εγώ πιστεύω κύριε Σιγητά ότι η έκκληση προς όλες τις πλευρές προς αυτή την κατεύθυνση είναι κάτι που πρέπει να προσθεθεί στην έκθεσή σας. Κατά τα άλλα συμφωνώ με την γενική κατεύθυνση που πάει η έκθεση, τη στηρίζω και προσβλέπω σε καλή συνεργασία με τον κύριο Χόβιτ προκειμένου να καταλήξουμε στο τελικό κείμενο της έκθεσης αυτής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η ε, κύριε Κορνέλισον έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Χόουιτ πρώτα απ' όλα για το τόσο καλό σχέδιο έκθεσης με τόσο πολλά καλά σημεία. Και την προηγούμενη φορά είχα μιλήσει για αυτή την έκθεση, είχα αναφερθεί στο μηχανισμό διατησία και χαίρομαι που τον βλέπω και τώρα εδώ. Και το σημείο 2 βέβαια πιστεύω ότι διατυπώνεται πάρα πολύ καλά αυτή τη φορά. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε δύο πράγματα κυρίω. Πρώτον, το θέμα του ονόματος. Έχουμε ετοιμάσει ένα κείμενο για τροπολογία που λέει ότι χαιρόμαστε για την πρωτοβουλία του Επιτρόπου Φίλε που θέλει να βάλει τους Πρωθυπουργού να συζητήσουν και να προχωρήσει η διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών με αυτόν τον τρόπο περισσότερο. Και αυτό γιατί πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβει κάποιο ρόλο προκειμένου να λυθεί το ζήτημα αυτό και επικοδομητικά να βοηθήσει. Άκουσα όμως ότι διαφωνεί η Ελλάδα με την πρόταση αυτή του κυρίου Φίλε. Δεν ξέρω, ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γνωρίζει περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Αν γνωρίζετε δηλαδή ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, αν όντω έτσι έχουν τα πράγματα. Επίσης πιστεύουμε ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εκφράσουμε μια σαφή δέσμευση για μια λογική λύση. Θα μπορούσαμε να παίξουμε ένα επικοδομητικό ρόλο, νομίζω, αν εμείς είμαστε ξεκαθαροί. Γι' αυτό και θα προτείνουμε να συμπεριλάβουμε το εξή. Χαίρεται για την πρόταση σύνθετου ονόματο με γεωγραφικό προσδιορισμό που προτείνει η ελληνική κυβέρνηση και πιστεύουμε ότι αυτό αποτελεί μια καλή βάση για συμβιβασμό εφόσον η ταυτότητα, η πολιτιστική γλώσσα κτλ. της Μακεδονίας δεν αμφισβητούνται. Τέλος. Για μας αυτή είναι η μόνη λογική λύση και πιστεύουμε ότι εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να το υποστηρίξουμε. Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι το θέμα των θεωρήσεων. Υπάρχει μια πρόταση εδώ που δεν είναι ξεκάθαρη. Λέει ότι το θέμα των Ρώμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να εμποδίζονται τα ταξίδια κλπ. Εγώ θα ήθελα εδώ να το διατυπώσουμε πιο ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει μηχανισμός άρσης προς το παρόν. Έτσι κι αλλιώς μπλοκάρει το διάλογος για άλλους λόγους. Αλλά θέλω να πω ότι είναι ένα πρόβλημα με πολλά πρόσωπα. Το θέμα είναι οι εθνικές μειονότητες να μπορούν και μέσα στη Σερβία και μέσα στη Μακεδονία να έχουν ένα λαμπρό μέλλον και όχι να θέλουν να ζητούν άσυλο. Συγχρόνως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι πιο ευάλωτοι θα πρέπει να προστατευτούν και όχι να γίνεται ακόμα χειρότερη η κατάστασή τους. Δεν τους βοηθάμε αν τους εμποδίζουμε να βγουν από τη χώρα επειδή δεν τους δίνουμε ας πούμε διαβατήριο. Πρέπει να προτίσουμε για αυτά τα ευάλωτα άτομα να έχουν καλύτερη κατάσταση μέσα στη χώρα. Κατά τα ευχαριστώ πολύ κύριε Χόβιτ. Ο κύριος Τάνοκ τώρα. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια στο Ρίτσαρντ ε, Χόβιτ. Και άλλη μια εξαίρετη έκθεση που ετοίμασε. Γι' αυτό το θέμα το οποίο έχει κρατήσει πολύ όσον αφορά την Μακεδονία και την ε, ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ και 8 χρόνια δεν τους επιτρέπουμε να αρχίσουν διαπραγματεύσεις εξαιτία του ζητήματος του ονόματος. Κατά τα άλλα η έκθεση μοιάζει με την προηγούμενη έκθεση. Η Μακεδονία λέει ε, προσπαθεί σκληρά, εγκρίνει όσο μπορεί περισσότερο από το ευρωπαϊκό κεκτημένο ως υποψήφια χώρα, χωρίς όμως να μπορεί να υπάρξει έναρξη επίσημα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Προφανώς έχει αποσταθεροποιηθεί πρόσφατα η Μακεδονία εξαιτία κάποιων δηλώσεων όχι πολύ σοφών από την Αλβανία όσον αφορά την ακαιρεότητα της δημοκρατίας της Μακεδονίας κάτι το οποίο βέβαια ανησυχεί την κυβέρνηση των Σκοπίων και είναι θλιβερό κατά τη γνώμη μου. Κατά τα άλλα η ομάδα μου στηρίζει την διαδικασία προσχώρησης και θέλει να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην αρχίζουν. Η Μακεδονία χρειάζεται ένα ιδιαίτερα θετικό μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ για να σταθεροποιηθεί η χώρα αυτή και να έχει αναγνωρισμένα διεθνώς σύνορα. Ελπίζω φέτος η ανησυχία από πλευρά τη Ελλάδα να έρθει και να μπορέσουν να αρχίσουν οι ενταξιακέ διαπραγματεύσει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προσωπικά είμαι υπέρ της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στην περιοχή των Βαλκανίων, αλλά θεωρώ ότι η διεύρυνση αυτή πρέπει να γίνει με σταθερά βήματα και να μην κυρονδοτήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τοπικά προβλήματα τα οποία είναι ανιστόρυτα. Ε, είναι γνωστό ότι υπάρχει διένεξη όχι μόνο σχετικά με το όνομα και επειδή ακούω ότι μόνο με το όνομα υπάρχει διένεξη με την Ελλάδα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το όνομα είναι όχημα αλλητρωτικών διαφορών τις οποίες εισάγει η Φύρομ κατά της Ελλάδος. Ήδη στη διαδρομή των πολλών ετών από τη στιγμή που το κράτος αυτό ε, ανεγνωρίστη η Ελλάδα έκανε πολλά βήματα προς τα πίσω. Πέρσι είχαμε μια συζήτηση με τον κύριο Χόιρη ως σκιώδης συγητής επί του θέματος. Ε, επέμενε στην άποψη ότι πρέπει να περάσουμε τον όρο Μακεδονικός και την οποία επαναλάβει και σήμερα ε, ελπίζοντας ότι θα έκανε τα βήματα τα οποία χρειαζόταν για να βρεθεί πιο κοντά με την Ελλάδα και τις λοιπές χώρες η Φύρο. Του είχα πει και πέρσι ότι αμφιβάλλω αν γίνει αυτό. Πέρασε ένας χρόνος, δεν έγινε κανένα βήμα. Πληροφορώ ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο εζήτησε συνάντηση και επαφή με τους αρμοδίους των Σκοπίων για το θέμα του ονόματος. Την όμως η απάντηση ήταν αρνητική. Με λυπεί λοιπόν το γεγονός ότι εκφράζει την ικανοποίηση του ο εισηγητής στο ζήτημα 9 εκφράζει τη λύπη του για, ότι το όνομα στέκεται εμπόδιο. Δεν είναι το όνομα που στέκεται εμπόδιο. Είναι η πίσω από το όνομα αλυτρωτισμή αυτού του κράτους το οποίο εμένα μου είναι συμπαθέστατο διότι αν θεωρούν ότι είναι Μακεδόνες είναι Έλληνες. Διότι γνωστόν της ιστορίας είναι ότι οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες. Με ενοχλεί βέβαια να υπάρχει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου καπηλευόμενων εις τα Σκόπια. Δεν με ενοχλεί να υπάρχει το άγαλμα του Λίτλ Αλεξανδρόφσκι εις τα Σκόπια. Του Σλάβιαν Αλεξανδρόφσκι. Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές με την Ελλάδα ε, ρίζες. Εάν τις θέλουν και επιθυμούν να έχουν τις ρίζες της Ελλάδος, ας μας το πούνε ευθέως και θα κοιτάξουμε να ε, ευπρόσδεκτα να τους δούμε σαν Έλληνες. Εάν προσπαθούν να αμφισβητήσουν τον ελληνικό μακεδονικό χαρακτήρα της ιστορίας, τότε εκεί είναι το πρόβλημα. Πιστεύω ότι όπως τα μικρά παιδιά επιμένουν σε ορισμένα πράγματα, το νεοσύστατο αυτοκράτος επιμένει σε κάτι το οποίο είναι αντίθετο και προς την ιστορία και δημιουργεί διανέξεις όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά και με τη Βουλγαρία. Συνεπώς, θα ήθελα να πω ότι η έκθεση και όλοι μας πρέπει να τα λάβουμε αυτά υπόψη. Δεν υπάρχει διένεξη εκ μέρους της Ελλάδος. Υπάρχει επιμονή και διένεξη εκ μέρους των Σκοπίων, της κυβερνήσεως των Σκοπίων. Και δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι το γεγονός ότι κάνουμε φιλοκυβερνητικές εκθέσεις, διότι η έκθεση είναι φιλοκυβερνητική προς το κυβερνητικό κόμμα. Δεν αποδίδει, διότι και την εσωτερική ένταση εξακολουθεί να την έχει. Είδατε από 24 Δεκεμβρίου η χώρα αυτή βρίσκεται σε μια έντονη εσωτερική πολιτική κατάσταση για διάφορους λόγους και ουσιαστικό αποτέλεσμα στην πρόοδο της ίδιας της χώρας της διεθνής της σχέσης δεν έχει. Συνεπώς, Εκείνο το οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι χρήσιμο και ωφέλιμο προς πάσαν κατεύθυνση είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί επιτέλους ποιο είναι το πρόβλημα. Ο ελληνικός λαός επιθυμεί να συμβιώσει. Δεν καταλαβαίνω οι άλλοι γιατί δεν επιθυμούν να συμβιώσουν με τον ελληνικό λαό και έχουν ε, βλέψεις εδαφικές. Ας κάνουν ρηματικές δηλώσεις σύμφωνες με το διεθνέ δίκαιο και να σταματήσει αυτή η ιστορία. Με συγχωρείτε που λέω ίσως παραπάνω κουβέντε, αλλά πρέπει να γίνει αντιληπτό το τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα των Βαλκανίων. Εμένα μου είναι συμπαθέστατη προσωπικά. Ω προ το θέμα, το ζήτημα του ονόματο θεωρώ ότι θα πρέπει να πάει όχι ως μεμονωμένο κεφάλαιο, αλλά σε υπό το κεφάλαιο σχέσεις καλής γειτονίας, περιφερειακή και ελληνική συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Uh, πολύ σύντομα να συγχαρώ τον κύριο Χάουιτ για την έκθεση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ολοκληρωμένη Προσωπικά, αλλά νομίζω και εξ ονόματος της ομάδας μου, αν και αυτή τη στιγμή είμαι μόνη εδώ, ούτως υπήν, νομίζω ότι πράγματι πρέπει να επιμείνουμε αυτά τα εκρεμή θέματα να λυθούν το ταχύτερο δυνατόν. Διότι μου φαίνεται ότι ενώ αφενός οι επαφές που αναφέρθηκαν και που προβλέπονται ή άρχισαν σε ανώτερα επίπεδα μεταξύ Μακεδονίας και, Ελλάδα, και Ελλάδας προετοιμάζονται, παράλληλα υπάρχει σκλήρινση των θέσεων ένθεν και κήθεν όπως ακούσαμε στη συζήτηση αυτή στο κοινοβούλιο μας. Αν συνεχιστεί αυτό θα επιδεινωθεί η κατάσταση. Και μου φαίνεται ότι όσο περισσότερο μένει απομονωμένη η Μακεδονία και διατηρεί αυτό τον προθάλαμο πιθανών ε, διαπραγματεύσεων, θα χειροτερέψει η κατάσταση και στη Μακεδονία, λέει η Μιλήτρια. Επιμένω λοιπόν να καταβληθούν προσπάθειες για την επίλυση του προβλήματος. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα ε, όπου έχουμε συνηθίσει να διαπραγματευόμαστε ημέν με τους δε και βέβαια ε, ξέρω ότι πολλές φορές τέτοιες καταστάσεις οδηγούν σε γελίες εξελίξεις. Μπορεί να τη συμβεί και αυτό. Εν προκειμένου όμως πρέπει να λυθεί το θέμα όσο γίνεται ε, γρηγορότερα και πρέπει και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να συμβάλλουμε στη λύση. Γιατί ωραία και καλά είναι να αναφέρονται οι δύο πλευρές σε ιστορικά στοιχεία που αν δεν κάνω λάθος λίγος πολύ έχουν ηλικία 2.000 ετών και βεβαίως όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα αλλά είναι αδύνατον πραγματικά δύο χώρες να αναγνωρίσουν ότι ένα, μια αξιόλογη προσωπικότητα που έζησε λίγο, γιατί πέθανε πολύ νέος, που έζησε πριν από 2.000 χρόνια, Δηλαδή δεν μπορεί να συμφωνήσουν ότι η προσωπικότητα αυτή ανήκουν και στις ιστορίες των δύο χωρών και δεν είναι μονοπόλιο μιας. Δηλαδή ε, στο πνεύμα του ευρωπαϊσμού θα πρέπει να είναι δυνατόν να συμφωνήσει κανείς πάνω σε μια τέτοια προσέγγιση. Ε, έκκληση λοιπόν προς όλους τους ενδιαφερομένους. Προσπαθήστε να βρείτε μια πρακτική λύση βιώσιμη αντί να πολλώνεστε και να σκληραίνετε τις αρχικές σας θέσεις. Ευχαριστώ. Bene, abbiamo concluso la lista degli shadow. Μάλιστα. Κλείσαμε τον κατάλογο των σκιωδών εισηγητών. Ε, μετά έχω ένα μακρύ κατάλογο συναδέλφων που θέλουν να πάρουν το λόγο. Πρώτη η κυρία Κοπά. Δύο λεπτά έκαστος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Χάουιτ για τη φετινή του έκθεση και θα πρέπει να πω πως συμφωνώ με τα όσα λέει για το πολιτικό κλίμα στην χώρα. ενώ η χώρα μπαίνει σε μια ε, χρονιά ύφεση με 21% ανεργία, διαπιστώνουμε και παρακολουθούμε μια σοβαρή πολιτική κρίση που εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παρακολουθήσουμε και να κρίνουμε αντικειμενικά. Επίσης πρέπει να εκφράσουμε ανησυχία για τις τελευταίες εξελίξεις και η Κομισιόν να δώσει μια αντικειμενική εικόνα στην έκθεση που θα παρουσιάσει την Άνοιξη. Σε αυτό το πλαίσιο οι υπερχόμενε εκλογέ είναι πάρα πολύ σημαντική δοκιμασία που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ε, προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ σε σχέση με τη θέση μας για τους διάφορους πολιτικούς, απέναντι στους διάφορους πολιτικούς φορείς και την κυβέρνηση. Γιατί θα ήταν μεγάλο σφάλμα να κρατήσουμε θέση ανάλογα με τις πολιτικές μας πεπιθήσεις, ένα λάθος που εμείς το Ευρωκοινοβούλιο συχνά κάνουμε. Να είμαστε λοιπόν ειλικρινείς και να βοηθήσουμε τις πλευρές να βρουν λύση. Ξέρουμε ότι η θέση μας είναι κατά των κενών εδρών στο Κοινοβούλιο, αλλά ας δούμε και για ποιο λόγο έχει δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση. Να μην κρατήσουμε λοιπόν κάποια θέση ανάλογα με την πολιτική μας κλίση. Δηλαδή, το αγαπημένο μου θέμα τώρα το όνομα. Στον, στην αξιότιμη συνάδελφο κυρία Νέτς, ναι, η ιστορία είναι για τους ιστορικούς. Όμως η, ε, ο Αλυτρωτισμός είναι για, τους, για εμάς, τους πολιτικούς και για αυτό το πράγμα μιλάμε εδώ. Ε, δώσαμε νέα όθηση στην ε, διαπραγματεύσεις και ε, η Ελλάδα στηρίζει και καλωσορίζει τις νέες πρωτοβουλίες ε, των πεσταλμένων που επισκέφθηκαν την Αθήνα και το Σκόπια την περασμένη εβδομάδα και έδωσαν νέες ιδέες, φρέσκες ιδέες. Ε, επίσης στηρίζουμε την προσήλωση του Επιτρόπου Φίλε. Θεωρούμε ότι έχει σοβαρό ρόλο να παίξει η Κομισιόν στο θέμα. Αλλά η δική μας συζήτηση, μια τελευταία λέξη. Η συζήτησή μας ε, για την Κροατία ε, ενίσχυσε τη θέση μα ότι τα διμερεί δήματα θα πρέπει να λύνονται όσο γίνεται πιο γρήγορα. Πριν καν την έναρξη διαπραγματεύσεων. Γιατί διαφορετικά θα είμαστε στην ίδια θέση που είμαστε τώρα. Δηλαδή να βρούμε ένα ενδεχόμενο πλάνο Β, όπω στην περίπτωση τη Κροατία. Και αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μα και να το κρατήσουμε ω δίδαγμα από τη συζήτηση περί Κροατία. Ο κύριο Κυρίλοφ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να σας ότι ο συγγετής δεν έχει εύκολη δουλειά. Προσπαθεί βέβαια να κάνει ό,τι καλύτερο. Έχει ήδη συμπεριλάβει βέβαια πολλά σημαντικά θέματα. Πρέπει να σας πω ότι η Βουλγαρία πάρα πολύ υπομονετικά περίμενε να λυθεί το ζήτημα του ονόματος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η τάση που υπάρχει εθνικισμού ε, την οποία βλέπουμε από τους γειτονές μας. Δεν έχει να κάνει μόνο με ιστορικά γεγονότα και όχι με 2.000 χρόνια πριν, αλλά και με πριν από λίγες δεκαετίες. Και τη δικιά μας, ε, η δικιά μας ιστορία χειραγωγείται, βλέπουμε. Προτείνεται, υπάρχει στο κείμενο και θα το υπογραμμίσει φαντάζομαι και ο Ρίτσαρτ, ότι εντάξει αφού δεν έχουμε να τα βάλουμε με την ιστορία, τουλάχιστον να γιορτάζουμε από κοινού κάποια ιστορικά γεγονότα. Τον Απρίλιο που μας πέρασε, εμείς πήγαμε να αποτιμήσουμε φόρο τιμής σε κάποιον από τους ήρωές μας που αντιστάθηκε στην τουρκική κατοχή και δέχτηκε επίθεση. Η αστυνομία δεν έχει βρει ακόμα τι έγινε. Ήταν πρέσβης, έτσι, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Άρα, τέτοιου είδους από κοινού γιορτασμοί, γιορτασμοί δεν λαμβάνουν χώρα. Αυτό που πρέπει συνεπώς να υπογραμμίσουμε είναι να προσπαθήσουμε να έχουμε καλές σχέσεις γειτονίας, η Μακεδονία δηλαδή, και με την Ελλάδα και με τη Βουλγαρία. Η Μακεδονία συμφώνησε να έχει διαπραγματεύσεις, έχουμε ομάδες εργασίας, αλλά θα υπάρξουν αποτελέσματα ή πρόκειται απλώς και μόνο για λόγια. Αν δούμε τι γίνεται με το ζήτημα του ονόματος, φοβούμαστε ότι και στη δικιά μα την περίπτωση μπορεί να μην προχωρήσουμε. Λοιπόν, πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε πραγματικά, να μην διονίζουμε. Θέλουμε να είμαστε επικοδομητικοί, αλλά συγχρόνως πρέπει να βάλουμε συγκεκριμένου όρου και προποθέσει. γιατί χωρί αυτού δεν μπορεί να υπάρξει καλό κλίμα ε, σχέσεων γειτονίας. Κάτι ακόμα εδώ. Η έκθεση αναφέρεται στο κόστος της μη διεύρυνσης. Είναι πολύ καλό που ο Ρίτσαρντ μας δίνει διάφορες ιδέες. Όσον αφορά λοιπόν τα τελευταία γεγονότα, η αντιπολίτευση άφησε το κοινοβούλιο. Άκουσα ότι Κάποιοι βουλευτές από την αντιπολίτευση έχουν συλληφθεί από την αστυνομία. Συμβαίνει κάτι τέτοιο, ισχύει. Ερώτηση είναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέει ο κύριος Κόβατσεφ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χόβιτ, για την πρότασή σας. Ελπίζω να καταλήξουμε σε κάποιο συμβιβασμό ώστε να μπορέσουν όλοι να τη στηρίξουν. Όλοι εδώ στηρίζουμε την ιδέα της ευρωπαϊκής ε, ολοκλήρωσης και της ένταξης της Μακεδονίας. Αλλά ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχουμε δεν είναι να σιωπούμε απέναντι στα προβλήματα. Αντίθετα, πρέπει να τα υπογραμμίζουμε, ιδιαίτερα εκείνα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Και εδώ αναφέρομαι στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου και τις ε, σχέσεις με τις γείτονες χώρες. Το πρόβλημα έχει να κάνει όχι με την ιστορία, αλλά με τις διακρίσεις που γίνονται σε βάρος πολιτών της χώρας, οι οποίοι μιλούν για την προέλευσή τους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την Βουλγαρία, όταν λένε ότι είναι Βούλγαροι δηλαδή. Και εδώ θα έπρεπε να υπάρξει κατανόηση. Και ρωτάω εδώ τους εκπροσώπους της Μακεδονίας, το αντιλαμβάνονται το πρόβλημα. Για άλλη μια φορά λοιπόν θέλω να κάνω έκκληση στα Σκόπια να, έρθει σε, να έρθουν σε επαφή με τους εκπροσώπους της βουλγαρικής κοινότητας ώστε να υπάρχουν συνεχείς επαφές και έτσι να ενημερωθούν, να μάθουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί. Τώρα θέλω να αναφερθώ στην νομοθεσία που έχει να κάνει με το άνοιγμα των αρχείων και παλιών υποθέσεων. Στην Επιτροπή αυτή που έχει δημιουργηθεί, υπάρχει επιρροή για δυσφήμιση κάποιων ατόμων και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με προηγούμενες προσπάθειες που έχουν γίνει στην Κεντρική και στην Ανατολική Ευρώπη για να ε, καταπολεμηθεί η κληρονομιά της κομμουνιστικής περίοδου. Τώρα εγώ θα επαναλάβω, για να τελειώσω, αυτά που είπαν και οι συνάδελφοι ότι προβλήματα υπάρχουν, υπάρχουν τα γεγονότα και πρέπει να δούμε τι γίνεται στο Κοινοβούλιο και τι γίνεται με τους ηγέτες της αντιπολίτευσης που ουσιαστικά εκδιώχθηκαν από τη Βουλή. Η ελευθερία έκφρασης αποτελεί στοιχείο κλειδί για μας. Πριν από λίγες μέρες ακούσαμε ότι είναι μερικό ελεύθερη χώρα η Μακεδονία. Οπότε να προσέξουμε πάρα πολύ όλα αυτά τα σοβαρά προβλήματα. Ευχαριστώ κύριε Σαγκουράκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να πω στον εισηγητή ότι συμφωνώ πάρα πολύ με το σημείο 25 τη έκθεσή του και ανησυχώ πάρα πολύ για την πραγματικά ψηλή ανεργία στην ε, γειτονική μα χώρα Απλά να σημειώσω όμως ότι αυτό το πρόβλημα έχει να κάνει με την όξυση της καπιταλιστικής κρίσης η οποία υπάρχει ούτως ή άλλως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ένταξη τη ε, της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση της κρίσης, της ανεργίας και της φτώχειας μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει. Δράτουμε τις ευκαιρία, να πω και στον κύριο Ρούτσεκ να πάει στους ε, συμπατριώτες τους, τους στην Τσεχία και να τους πει να ζήσουν με 100 ευρώ που είναι το αποτέλεσμα 20 χρόνων μεταρρυθμίσεων, κύριο Ρούτσεκ. Δεν είναι ότι στην Ελλάδα δεν υπήρχαν μεταρρυθμίσει, στην, στην Πορτογαλία ή στην Ισπανία. Υπήρχαν μεταρρυθμίσει και το αποτέλεσμα το ζούμε. 30% ανεργία και πολύ ψηλή ανεργία για του νέου. Γι' αυτό τα μαθήματα αλλού. Τώρα, για την έκθεση που μα αφορά. Ε, καταρχήν, ε, συγχαίρω τον κύριο Χάουιτ για το ότι ε, ασχολείται με το πρόβλημα της ανεργία. Βέβαια, αυτό που συστήνει ω λύση δεν είναι λύση διότι το πρόβλημα δεν θα λυθεί με κοινωνικό διάλογο, το πρόβλημα θα λυθεί με ανάπτυξη. Και όσο έχουμε καπιταλιστική σχέσει παραγωγή, ανάπτυξη δεν θα υπάρχει. Γι' αυτό το λόγο κιόλα, στην έκθεση φέτο, κύριε Χάουιτ και ούτε στην περσινή σα, δεν λέτε ποιο πρέπει να είναι το αναπτυξιακό πρότυπο αυτή τη χώρα. Τι πρέπει να παράγει η γειτονική χώρα για να λύσει τα προβλήματά τη. Επίση, θα πω κάτι γενικότερο, δεν αφορά μόνο την έκθεσή σα. Αλλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση όταν συζητάμε αυτέ τι εκθέσει δεν αναφερόμαστε σε προηγούμενε εκθέσει του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά αναφερόμαστε στο Συμβούλιο. Τέλο, ο μηχανισμό που προτείνεται στο σημείο 10, θα σα πω κύριο Χάουιτ ότι είναι προ σε βάρο τη γειτονική χώρα. Διότι όπω πολύ καλά είπε ο κύριο Πρόεδρο, όποιο μπήκε στο λεωφορείο θα προσπαθεί να εμποδίσει να μπουν άλλοι στο λεωφορείο. Γι' αυτό πρέπει να απαντηθεί ποια είναι η βάση επίλυση τέτοιων ζητημάτων. Θα είναι το διεθνές δίκαιο θα είναι ο ΙΕ ή θα είναι το δίκαιο του ισχυρότερου. Και το σημείο 10 εισάγει ακριβώς το, το δίκαιο του ισχυρότερου. Αυτό θα είναι σε βάρος και της γειτονικής χώρας και της Ελλάδας. Και εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει μια απάντηση γιατί δεν έχουν αποδώσει μέχρι τώρα τα ε, προσπάθειες το Αμερικανών Νίμιτς. Δεν ασχολείται με το θέμα του ονόματος. Τι παραπάνω θα προσφέρει ο, ο, ο κύριος Φίλε στο ζήτημα αυτό. Κυρία Γιαννάκου. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χόουτ για την έκθεσή του, η οποία βέβαια διαφέρει από την περσινή κατά το μέγεθος. Η περσινή έκθεση είχε 66 παραγράφους, η φετινή έκθεση έχει 24. Ε, αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κακό, ωστόσο έχουν παραλυφθεί ορισμένα ζητήματα που αφορούν στην εσωτερική κατάσταση της χώρας. Ε, δεν γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα γεγονότα της 24ης Δεκεμβρίου, τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Και βέβαια επαναλαμβάνεται η θεώρηση, η οποία αναφέρθηκε και εδώ από πολλούς συναδέλφους ως προς το όνομα. Δεν είναι το θέμα του ονόματος, κύριε Πρόεδρε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ ε, είναι άλλες ιστορίες οι οποίες δημιουργούνται. Είναι κυρίως αυτή η προσπάθεια αρχαιοποίησης των σημερινών προβλημάτων και αναζήτησης μιας ταυτότητας που δεν υπάρχει. Η Ελλάδα έχει κάνει συγκεκριμένα βήματα και μάλιστα το τελευταίο διάστημα ο Υπουργός Εξωτερικών απέστειλε μια επιστολή στον Υπουργό Εξωτερικών ε, της χώρας αυτής ε, ζητώντας να γίνει ένα memorandum of understanding και να αρχίσει από αυτό μια διαδικασία η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στη λύση του προβλήματος. Επίσης ο κύριος Νίμιτς επανήλθε, διότι η διαδικασία αυτή ε, γίνεται υπό, την, ε, υπό τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δεν είναι διμερές πρόβλημα το πρόβλημα της, ε, της ΦΥΡΟΜ, κύριε Πρόεδρε. Είναι διεθνές πρόβλημα. Δεν είναι διμερές. Και επομένως ασχολούνται με, ασχολούνται με αυτό τα Ηνωμένα Έθνη και ήρθε στην Αθήνα απογοητευμένο. Διότι όταν μια χώρα επενδύει σε μια ψεύτικη ε, ταυτότητα και αρχαιοποίηση, μετά βεβαίω αντιλαμβάνεστε ότι δυσκολεύουν τα πράγματα για να πείσει του ανθρώπους του οποίους έχει διδάξει πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Και βέβαια τα προβλήματα αυτά δεν είναι μόνο αρχαία προβλήματα. Είναι προβλήματα που έχουν σχέση με την ε, με τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και με την επιχείρηση η οποία έγινε να αποσπαστεί τμήμα της Ελλάδος. Επομένως, όταν το κυβερνόν κόμμα αυτή τη στιγμή στη χώρα αυτή ε, έχει ως τίτλο το «Ελεύθερη Μακεδονία» και το χάρτη όπου η Θεσσαλονίκη, η οποία ανήκει στην Ελλάδα, παρουσιάζεται ως πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Αυτά, συγχωρήστε με, είναι επίοικος κομικά. Δεν θέλει η χώρα αυτή πραγματικά κατά τη γνώμη μου να υπάρξει λύση για λόγους δικούς της. Mr. Posselt. Κύριος Πόσελτ, ευχαριστώ πολύ. Δύο θέματα. Πρώτον, συμφωνώ με την ε, λογική πρόταση Howitt που προσπαθεί και τη δύσκολη εσωτερική πολιτική κατάσταση στη Μακεδονία να την αξιολογήσει αντικειμενικά, όπως άλλωστε και ο Επίτροπος Φίλε. Και το είπα και στα μακεδονικά μέσα και στα κόμματα εκεί της Μακεδονίας ότι πρέπει να δουν το παράδειγμα των γειτονικών χωρών που προχώρησαν στο δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί η αντιπολίτευση δέχτηκε ότι η πλειοψηφία είναι δεδομένη, έχει μια πλειοψηφία τέλο πάντων και ότι θα περιμένουν μέχρι την ε, επόμενη θητεία για να αλλάξουν τα εκλογικά αποτελέσματα. Και στην πλειοψηφία λέω ότι η μειοψηφία έχει δικαιώματα και εκείνη. Αυτά λειτουργούν στη Μακεδονία καλύτερα από ό,τι φαίνεται αλλά θα πρέπει να αλλάξουν πολιτική. Ο Χέρμπερτ Βένερ, ένας παλιός Γερμανός πολιτικός που έφυγε από το κοινοβούλιο για λίγες ώρες, είπε ότι όποιος φεύγει πρέπει να μπορεί να ξαναγυρίζει. Και αυτό το ότι θα υπάρξει ε, μποϊκοτάρισμα της αντιπολίτευσης δεν ισχύει, όλοι πρέπει να συνεργάζονται. Τέλος, θα πρέπει να σταματήσουμε να ε, φέρνουμε στο προσκήνιο φαντάσματα. Άλλαξε το Σύνταγμα στο, στη Μακεδονία και στην αλλαγή αναφέρεται ότι δεν έχουν αξιώσεις από τις ε, γειτονικέ χώρες. Αλλιώς ε, θα ήταν πραγματικά αστεία η κατάσταση. Άλλαξαν όμως το σύστημα και ένα αντικείμενο της συμφωνίας ήταν η επίλυση και του ονόματος και άλλαξαν το ύμνο, το Σύνταγμα στη Μακεδονία και ακόμα μετά από κοντά 20 χρόνια εξακολουθεί να υφίσταται ως λόγος αποκλεισμού το όνομα. Εγώ είμαι υπέρ της προσέγγισης του Επιτρόπου Φίλ. Πρέπει να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις που έτσι κι θα πάρουν 8 με 10 χρόνια για να λυθούν όλα τα ερωτήματα, αλλά να αξιοποιήσουμε τον αποκλεισμό και να παρεμποδίσουμε τις διαπραγματεύσεις, αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Ευχαριστώ κύριε Πόσελτ. Και τώρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κύριος Ντέιβιτ Κάλνεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επανέρχομαι στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου που είναι σημαντικά γιατί ο εμφύρωμα είναι προορατικά, δεν είναι στατικά, όπως εκείνα των προηγουμένων ετών. Και μετά τα συμπεράσματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να δουλεύει για να προετοιμάζει την ερηνή έκθεση που ανατέθηκε από το Συμβούλιο και εξέτασε τρία θέματα. Τη συνεχιζόμενη υλοποίηση των προτεραιοτήτων στο διάλογο υψηλού επίπεδου για την προσχώρηση, την πρόοδο στις καλές, σχέσεις καλές γειτονίας, και βήματα για το, την επίλυση του ονόματος. Όπως ξέρετε, είναι λίγος ο χρόνος. Η προθεσή μας και η ελπίδα μας είναι να εγκριθεί μια έκθεση κάποια στιγμή τον Απρίλιο και αυτό σημαίνει ότι είναι σημαντικό να αρχίσουμε αμέσως να εργαζόμεθα. Έτσι λοιπόν ο Επίτροπος Φίλε ήρθε σε επαφή με όλους τους ομολόγους του και έστειλε αριθμό επιστολών καλώντας σε στενότερες επαφές και συντονισμό, διμερείς επαφές και τριμερείς επίσης. Αυτό που είναι σημαντικό εδώ είναι ότι η επαφές πρέπει να είναι ουσιαστικές, πρέπει να προσανατολίζεται προς τα αποτελέσματα και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις εξελίξεις, τις συνεχιζόμενες ε, συνεδριάσεις ε, που θα στοχεύουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα. Όλα αυτά θα τα αποτιμήσουμε σε το χρόνο. Τώρα για την πολιτική κρίση δύο λόγια, την οποία παρακολουθούμε πολύ από κοντά τι έγινε στις 24 Δεκεμβρίου και πριν είναι ανησυχητικό. Ο Γενικός Διευθυντής μας Ανίνο επισκέφθηκε την περασμένη εβδομάδα τη χώρα στα πλαίσια τακτικής συνεδρίασης και follow-up για την προετοιμασία της έκθεσης της Άνοιξης. Επίσης συνήντησε όλα τα μέρη για να, να συζητήσουν για την κρίση και τρόπους για να ξεπεραστεί το παρόν αδιέξοδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είχε την περασμένη εβδομάδα ε, συνάντηση με τον πρέσβη και ε, κάλεσε όλα τα μέρη να καλέσουν τις, τους θεσμούς, τις διαδικασίες και δημοκρατικές αξίες επί των οποίων εδράζεται το Κοινοβούλιο και κάλεσε το κόμμα της αντιπολίτευσης να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο. Εμείς ε, παρακολουθούμε, όπως βλέπετε, τις εξελίξεις ε, από πολύ κοντά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν συνόλο και σε επίπεδο διαλόγου υψηλού επίπεδου για την ε, προσέγγιση προβλέπεται επίσκεψη του Επιτρόπου σύντομα. Θα συνεχίσουμε τις προετοιμασίες μας για την έκθεση την Ερηνή και οι αρχές στα Σκόπια λαμβάνουν σειρά μέτρων σε όλους τους τομείς και τώρα μάλιστα ο Υπουργό Εξωτερικών Παπάσχη έχει συνάντηση με τον Επίτροπο Φίλε για να συζητήσουν τα μέτρα της κυβέρνησης ή μέτρα που προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση. Επίσης, ε, στα πλαίσια αυτά θα παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυ στη κατάσταση και όπως είπα θα ε, επιστρέψουμε στα Σκόπια σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σαλαβράκο, για διαδικαστικό ζητείτε το λόγο. Υπενθυμίσω στο σώμα ότι η Ελλάδα ήταν ε, το ένα από τα δέκα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έφερε αντίρρηση για την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα έχει 27 και άλλους υπό ένταξη. Δεύτερον, αφού το ανεφεί το θέμα υπάρχουν έξι κυβερνήσεις διαφόρων κομματικών σχηματισμών στην Ελλάδα ενώ ο ίδιος ε, κομματικός σχηματισμός κυβερνά τα Σκόπια από τις ιδρύσεώς τους, το ΒΜΡΟ. Ποτέ η Ελλάδα, τρίτον, δεν έχει απειλήσει, δεν έχει εκφράσει απειλή για τα Σκόπια. Και τέταρτον, πρέπει να, αντιληφθείτε ότι έχει πολλά σοβαρά προβλήματα η Ελλάδα και αυτό πρέπει, θέλει να το λύσει. Το γράμμα λοιπόν πρέπει να πάει στην διεύθυνση Σκόπια. This is not a point of order. Δεν ήταν διαδικαστικό. Τώρα, κύριε Χόβιτ, έχετε το λόγο για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Θα απαντήσω σε όλους. Ο κύριος Κούκαν και, ο κύριος, και η κυρία Κορνέλησο και η κυρία Γιαννάκου και ο κύριος Πόστο αναφέρθηκαν στο ίδιο θέμα. Θα πρέπει στην έκθεσή μας να λέμε κάτι για τα προβλήματα μεταξύ των πολιτικών κομμάτων όπως είπαν οι συνάδελφοι, πριν από τις 24 Δεκεμβρίου τίμασα εγώ την εκθεσή μου και γι' αυτό δεν αναφέρεται τίποτα για αυτά που είπατε. Ευχαρίστως μαζί σας να βρούμε τη σωστή διατύπωση και να το συμπεριλάβουμε. Ε, ξέρω τη δήλωση των ΗΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ισορροπημένες οι δηλώσεις και ίσως θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε αυτές ως σημείο κίνησης. Ε, για αυτό που είπε η κυρία Κορνέλισον τώρα, για κάτι πιο συγκεκριμένο όσον αφορά τη λύση στο ζήτημα του ονόματος. Όντως πρέπει να υπάρξει πυθός. Πρέπει να είμαστε σίγουροι για το ποια θα πρέπει να είναι η αποτελεσματική λύση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι θέλετε να βοηθήσετε, αλλά πρέπει να με πείσετε. Για το θέμα των θεωρήσεων, πιστεύω κι εγώ, όπως λέτε, ότι δεν είναι τόσο σαφές εκεί το θέμα. Συμφωνώ μαζί σας και εγώ όταν το ξαναδιάβασα αυτό σκέφτηκα. Αλλά η πρόθεσή μου είναι ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι Ρώμα ώστε να οδηγούμαστε σε διακρίσεις. το έχουμε συζητήσει ξανά και εδώ στις Βρυξέλλες ότι μερικές φορές ε, χρησιμοποιούμε άλοθη και περιορίζουμε το δικαίωμα στα ταξίδια. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τάνοκ, ιδιαίτερα για αυτό που είπε για την Αλβανία, γιατί για αυτούς που πιστεύουν ότι αυτή η χώρα μπορεί να παραμείνει στη θέση της και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει, το θέμα της δήλωσης της Αλβανίας δείχνει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αν θέλουμε λοιπόν ησυχία, ειρήνη και δημοκρατία στην περιοχή, σε όλες τις χώρες της περιοχής, δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή την χώρα απομονωμένη. Οπότε συμφωνώ μαζί σας. Στον κύριο Σαλαβράκο. λέει ότι προσωπικά συμπαθεί τη χώρα και κατανοεί και είναι υπέρ της διεύρυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία, να το βάλουμε αυτό στο κείμενο. Μεταφράστε αυτά που λέτε, δώστε μου μια διατύπωση να τη βάλουμε στο κείμενο. Όταν λέτε ότι δεν γίνονται βήματα προς τα μπρος, είπαμε ποια είναι αυτά που έχουν γίνει. Έχουν γίνει για το καθεστώς, Υπάρχουν ε, απαντήσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Και έχει υπάρξει η ανταλλαγή επιστολών με την Ελλάδα. Δεν συμφωνώ μαζί σας. Αλλά να συνεργαστούμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα κοινό τόπο. Κυρία Νέης, μπορεί να νιώθετε μόνη, αλλά εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι η χώρα να μην νιώθει μόνη, να μην είναι μόνη. Και στην κυρία Κοπά τώρα αλυτρωτικά. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι είναι μια χώρα η οποία, ε, μάλλον ότι έχει βλέψει προς μια χώρα η οποία πολιτικά ελέγχεται από κάποια άλλη. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Νέη σε αυτό. Ότι και οι δύο χώρες μπορούν να μοιράζονται μια κοινή κληρονομιά και ότι έτσι θα έπρεπε να λυθεί το θέμα. Ίσως να μην ήταν η πρόθεσή σας, αλλά το λέω γιατί δεν μπορεί να υπάρξει αλλιώς ακαιρεότητα κληρονομική. Συμφωνώ όμως με πολλά από αυτά που είπατε και προσπαθώ γενικά να συνομώ μαζί σας όσο γίνεται περισσότερο. Στον κύριο Κυρίλοφ. Τα... Οι κοινοί εορτασμοί, ναι, όλοι συμφωνούμε, αλλά τελικά γιατί ορτασμούς μιλάμε. Και εκεί είναι η δυσκολία το να αποφασίσουμε για ποιου εορτασμού μιλάμε, πώς θα συμφωνήσουν οι χώρες. Αλλά μακάρι αν μπορώ να βοηθήσω να υπάρχει διάλογος για να βρεθούν αυτοί οι κοινοί εορτασμοί, βεβαίω. Συμφωνώ με αυτό που είπατε για τις ομάδες εργασίας που δημιουργήθηκαν. Και τώρα για τις συλλήψεις της αντιπολίτευσης εγώ δεν παρεμβαίνω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Δεν ξέρω εσείς τι έχετε μάθει, εγώ δεν έχω πάντως τις ίδιες πληροφορίες. Κύριε Κόρβατσοφ, ευχαρίστως να έχουμε διάλογο και με άλλους συναδέρφους για να βρούμε τους σωστούς συμβιβασμούς. Και πέρυσι, για τις παραβιάσεις που έγιναν, εμείς πρέπει να ζητήσουμε διαφάνεια για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο χειρισμός δεν θα πρέπει να στοχεύονται άτομα. Ποτέ, από κανένα πολιτικό φάσμα. Νομίζω ότι συμφωνείτε μαζί μου. Στον κύριο Γκουράκη τώρα. Για το οικονομικό μοντέλο. Άκουσα ότι υπάρχουν σουηδικές και βρετανικές επενδύσεις. Οι μεταφορές θα υποφεληθούν, η βιομηχανία είναι μια υπέροχη χώρα για τον τουρισμό και εκεί υπάρχει τεράστιο δυναμικό. Οπότε να πιούμε ένα κρασί μαζί που προέρχεται από τη χώρα και που είναι νοστιμότατο. Αν όμως περιμένετε να λύσω εγώ τα προβλήματα του καπιταλισμού, φοβάμαι ότι εδώ θα διαφωνήσω. Έτσι κι είναι δύσκολο να προχωρούν οι συνομιλίε. Εγώ αυτό θέλω, για τα υπόλοιπα δεν μπορώ. Α το πετύχουμε αυτό και μετά βλέπουμε για τα υπόλοιπα. Κύριε Γιαννάκου, αναφέρθηκα νομίζω στι παρατηρήσει σας, ε, του κύριο Πόσελτ επίση, οπότε να τελειώσω με το εξή πρόεδρε. Είπα ήδη ότι τα δύο κύρια πολιτικά κόμματα έχουν ε, διάλογο σήμερα. Κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό. Να τον αγνωρίσουμε. Δείχνει ότι μπορούν να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Οι πληροφορίε που έχω εγώ, αλλά βέβαια είναι και αυτό που είπε η κυρία Κορνέλισον, είναι ότι δεν έχει απορρίψει τις συνομιλίες που προτείνω φίλε η Ελλάδα. Τώρα με την, ε, τον επόμενο γύρο θα δούμε. Ο Υπουργός Εξωτερικών, πάντως της, ο εκπρόσωπος μάλλον του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας είπε ότι δεν πρέπει να γίνονται συναντήσει αν δεν υπάρχει καλή προετοιμασία και δεν διασφαλίζονται ουσιαστικά αποτελέσματα. Άρα δεν υπάρχει απόρριψη. Και από αυτό που είπε ο κύριος Κρεύσκη, είπε μετά από τη δήλωση αυτή ότι θα συνεχίσουμε με θετικές κινήσεις γιατί εμείς θέλουμε το πρόβλημα αυτό να λυθεί. Και συνεχίζει εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα αναλυφθούν περισσότερες πρωτοβουλίες από διάφορες πλευρές και όσο αφορά εμάς πάντα είχαμε πρωτοβουλίες, ε, πίστη και διάθεση να λυθεί το πρόβλημα. Δεν υποτιμάω βέβαια τις διαφορές που υπάρχουν, αλλά όταν εκείνος ζητάει πρωτοβουλίες, ο τρόπος με τον οποίο εμεί το συζητάμε και πώς θα ψηφίσουμε το κείμενό μας είναι ήδη μια πρωτοβουλία. Και εγώ είμαι αποφασισμένος μέχρι τον Ιούνιο φέτος να έχουμε βρει τις προϋποθέσεις ώστε να αρχίσουν οι συνομιλίες και κάνω έκκληση στους συναδέρφους από όποια πολιτική πλευρά και αν έρχονται να συμφωνήσουν μαζί μου και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να το πετύχουμε αυτό. Σας ευχαριστώ. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 28 Ιανουαρίου, στις 6 το απόγευμα. Επόμενο σημείο. Ναι, 28, 28, συγγνώμη αν δεν με καταλάβατε. Περνάμε στο επόμενο σημείο, έκθεση πρόοδου 2012 για τη Σερβία. Ο εισηγητής είναι ο Γέλκο και όχι Τζέλκο Κάτσιν. Δεύτερη εξέταση του σχεδίου έκθεσης για τη Σερβία, που παρουσιάστηκε στην Επιτροπή στις 3 Δεκεμβρίου. Προθεσμία για υποβολή τροπολογιών ήταν η 9η Ιανουαρίου και υποβλήθηκαν 190 τροπολογίες. Δίνω αμέσως το λόγο στον εισηγητή κύριο Κάτσιν. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριε εκπρόσωπε της Επιτροπής, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδες εισηγητές και τους άλλους συναδέλφους για τις επικοδομητικές τους τροποποιήσεις. Είμαι ευτυχής διότι οι περισσότερες τροπολογίες ήταν σύμφωνες με το αρχικό μου σχέδιο. Όλες οι πολιτικές ομάδες συμφωνούν για τα κεντρικά ζητήματα και το πολιτικό μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε στους εταίρους μας στο Βελιγράδι. Ιδιαίτερα θα ήθελα να καλωσορίσω τις τροπολογίες του ΕΛΚΑ για το θέμα της Βοηβοντίνας και τις τροπολογίες για περιβαλλοντικές προκλήσεις που υπέβαλαν οι πράσινοι. Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για συμβιβαστικές τροπολογίες που θα είναι έτοιμες μέχρι την Πέμπτη. Σε σχέση με τα βασικά τη βασική προτεραιότητα του κοσμοπεδίου υπήρξε κάποια πρόοδος από την πρώτη εξέταση της έκθεσης αυτής της ε, 3 ε, Δεκεμβρίου. Ο Πρωθυπουργό Ντάτσης της Σερβίας έκανε έναν πρώτο γύρο ε, συζητήσεων με τον ε, ομόλογό του την περασμένη εβδομάδα έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις σχέσεις της χώρας με το κοσμοπέδιο. Τον έφερε και χτες όταν συζητήσαμε το ε, Κωσυφοπαίδιο. Τη συμφωνία λοιπόν ε, θα πρέπει να επεκταθεί σε όλες ε, τις συνοριακές διαβάσεις. Η εφαρμογή των υπολείπων συμφωνιών εξελίσσεται ομαλά. Το θέμα είναι το Βόρειο Κωσυφοπαίδιο, που το ψήφισμα ασχολείται λεπτομερώς με αυτό το θέμα. Καθιστάμε σαφές ότι διχασμός του κοσυφοπεδίου με βάση εθνοτικά ζητήματα δεν θα είναι δυνατή. Ως προς αυτό, λοιπόν, θα πρέπει να υιοθετηθεί το ψήφισμα του διαλόγου που υιοθετήθηκε στην Πρίστινα τον Ιανουάριο. Ε, εδώ θεμεσμοθετείται και νομοποιείται ο διάλογο, υπογραμμίζονται οι προτεραιότητε και υπογραμμίζεται η σημασία τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση τη Σερβία και τη περιφέρεια. Εγώ διαφωνώ με τις ερμηνείες γιατί ο κύριος Πόσελτ είπε κάτι της προάλλες σε σχέση με το ψήφισμα το οποίο καλούμε να εκτιμήσουμε τις θετικέ του πτυχέ και επιπτώσεις. Εγώ πιστεύω ότι είναι σημαντικό βήμα μπροστά σε σχέση με την προηγούμενη Ε, λύση. Για το Πρέσοβο, Μπουγιάνοβας και Μέτζεβα και για τον εορτασμό της, ε, των ηρώων που έπεσαν στις ε, μάχες σε αυτά τα μέρη και στο μνημείο που απομακρύνθηκε το Κυριακή δεν υπήρξαν εκεί προβλήματα. Ωστόσο θα ήθελα να καλέσω τους, ε, όλες τις πλευρές ε, να προσπαθήσουν ε, να κατευνάσουν τα πνεύματα. Για τους Αλβανούς θα πρέπει να γίνουν περισσότεροι, περισσότερα πράγματα, οι Σέρβοι να τους δεχτούν και οι Αλβανοί ηγέτες της περιοχής να κάνουν προσπάθειες. Δυστυχώς όμως βεβηλώθηκαν τάφοι και, και, και κλεισίες στο Κωσυφοπαίδιο ανάμεσα στην Κυριακή και στη Δευτέρα. Εγώ Καταδικάζω αυτή τη βία και ελπίζω πως οι αρχές του Κωσυφοπεδίου θα εμποδίσουν ε, την επανάληψη τέτοιων επεισοδίων. Ε. Αυτοί που προέβησαν σε αυτές τις ευέβλε πράξεις θα πρέπει να, καταδικα... να συλληφθούν και να δικα... καταδικαστούν. Ε. ο σεβασμός της ανεξιδρυσκείας είναι δικαίωμα και απόδειξη κάθε πολιτισμού. Ε, πολιτισμένης χώρας. Θα πρέπει λοιπόν οι αρχές της χώρας να εξασφαλίσουν το σεβασμό αυτών των δικαιωμάτων για όλους προς χάρη των νεότερων γενεών και προς χάρη του ευρωπαϊκού τους μέλλοντος. Να ε, ε, καλωσορίσω τη συνάντηση του Τάτζης και Μιλάνοβιτς Πρωθυπουργών Σερβίας και Κροατίας στη... που οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι σημαντικές για ολόκληρη την περιφέρεια και η πολιτική και η οικονομική συνεργασία μπορεί να βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό. Από την άλλη πλευρά, η καταπολέμηση συστηματικής διαφθοράς περνά σε μια επόμενη φάση ο αναπληρωτής Πρωθυπουργό Βούτση σε αυτή την ε, προσπάθεια έχει δώσει νέα δυναμική στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στην αλλαγή της σερβικής πολιτικής εν γέννη. Θα πρέπει να καλωσορίσουμε αυτή τη διαδικασία και να θαρρύνουμε τους Σέρβους ηγέτες να, ε, εντατικοποιήσουν αυτές τις ε, προσπάθειες καταπολεμώντας τη διαφθορά στις δημόσιες επιχειρήσεις που ελέγχονται από τα πολιτικά κόμματα στη Σερβία. Ταυτόχρονα μόνο η καταπολέμηση τη δεν πρέπει να γίνεται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανακοινώντα τι μελλοντικέ δράσεις. Αυτή η πρακτική βαθμίζει, υπονομεύει το κράτος δικαίου στη χώρα και πρέπει να πάψει. Το ίδιο σημαντική είναι η δουλειά των ανεξάρτητων ρυθμιστικών σωμάτων, όπως οι κρατικές υπηρεσίες ελέγχου, οικονομικού ελέγχου, που πρέπει να έχουν την οικονομικές και διοικητικές ε, πηγές, γιατί μόνο ισχυρά και ανεξάρτητα θεσμικά όργανα θα έχουν αποτελέσματα στην καταπολέμηση της διαφθοράς ε, και μόνιμα αποτελέσματα. Να τονίσω το θέμα της άσχημης οικονομικής κατάστασης της χώρα. Η ανεργία φτάνει το 27%, η ευτόχεια αυξάνεται, ενώ η στριμωγμένη μεσαία τάξη δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Επενδυτές διστάζουν να επενδύσουν στη Σερβία από τη στιγμή που έχουν να αντιμετωπίσουν τόσε αβεβαιότητε. Γι' Η καταπολέμηση της διαφθοράς θα πρέπει να συμβαδίζει με τη δημιουργία ανεξάρτητων θεσμών και επαγγελματικού δικαστικού σώματος. Σε τρεις μήνες από τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναφερθεί στην Κομισιόν, στο Συμβούλιο, με για την πρόοδο στο, στη, της Σερβίας. Εγώ πιστεύω πως η Σερβία θα ενεργήσει υπεύθυνα και ότι σε το χρόνο τα εκρεμή ζητήματα θα ρυθμιστούν έτσι ώστε το Συμβούλιο να είναι σε, θέμα, σε θέση να ορίσει την ημερομηνία για την έναρξη των ε, μεταξιακών διαπραγματεύσεων. Προσβλέπω σε αυτή την ημερομηνία όταν δηλαδή η Σερβία θα μπει, θα ανέβει στο τρένο ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, προσβλέπω στη συζήτηση για αυτή τη δεύτερη εξέταση της έκθεσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κατσίν. Ο κύριος Σλέφλιν, σκιώδης εισηγητής του ΕΛΚ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στον Γέλκο Κατσίν για την καλή έκθεση που είναι και είναι και φόρος τιμής ε, για την ποιότητα, οι 190 τροπολογίες, ε, εκ των οποίων πολλές ε, ταιριάζουν με το ύφος της έκθεσης. Δεν θα μπω στην ουσία, όπως είπε και ο κύριος Κατσίν και σε προηγούμενες συζητήσεις τέθηκαν θέματα και από τον ίδιο και από άλλους. Τρεις παρατηρήσεις. Μια ιδέα του κυρίου Χάουτ που κρίμα που έφυγε γιατί είναι ενδιαφέρουσα η ιδέα Δηλαδή ότι κάθε χώρα πρέπει να αφήνει ένα κομμάτι του ΑΕΠ της για τους ΟΤΑ και την περιφερειακή και τοπική κυβέρνηση. Αυτό είναι σημαντικό, όχι για αυτή την έκθεση φέτος, αλλά για επόμενες. Ας το κρατήσουμε. Δεύτερον και σοβαρότερο ένα θέμα που έθεσα σε προηγούμενη συζήτηση, το Σύνταγμα της Σερβίας που είναι ένα πρόβλημα. Δηλώνει ότι το κοσυφοπαίδιο είναι οργανικό κομμάτι της εδαφική επικράτειας της Σερβία. Αυτό πρέπει να αλλάξει, δεν γίνεται να μείνει, γιατί στο βαθμό που το δεχόμαστε θα δεχτούμε και ότι υπάρχει μια νομική αντίφαση στην καρδιά της διαδικασίας που ε, προωθούμε. Δηλαδή την ε, κάποια στιγμή την προσχώρηση της Σερβίας. Η Σερβία και το Κωσυφοπέδιο δεν είναι προβλήματα που θα εξαφανιστούν ακόμα κι αν λυθούν όλα, ακόμα κι αν επικρατήσει η ειρήνη και πέφτει ο ένας στην αγκαλιά του άλλου μέσα σε κλίμα αγάπης και αλληλεγγύης. Το πρόβλημα είναι ότι η Σερβία θα εξακολουθεί να είναι γειτονική, συγγενική χώρα του στο Κωσυφοπέδιο στο βαθμό που θα υπάρχει σερβικός πληθυσμός στην τελευταία θα υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει σχέση πάντα μεταξύ Σερβίας και Σέρβων του Παιδίου. Είναι η κοινότητα μεγάλη και δεν εξαφανίζεται η σερβική κοινότητα. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά είναι το εξή. Οι Σέρβοι του Παιδίου δεν δέχτηκαν να γίνουν πολίτες του Παιδίου. Αυτή η διαδικασία όπου δόθηκαν στο Παιδίου γίνεται για να διασφαλιστή ενότητα. Αυτό πρέπει να το υποστηρίξουμε και η υπόσταση του κράτους για την εσωτερική σταθερότητα του Κωσυφοπεδίου και για τις σχέσεις με τη Σερβία. Ε, όλοι αυτοί οι παράγοντες θα εξακολουθήσουν να παίζουν ρόλο. Ο κύριος Ρούτσεκ πριν με είπε ε, απεσιόδοξο. Αν και είμαι Ούγγρος, δεν είμαι απεσιόδοξος, είμαι ρεαλιστής. Και μέσα από αυτό το πρίσμα πρέπει να δούμε και ένα άλλο πιθανό σενάριο, πιθανό, αλλά συζητείτε και στα Τύρανα και στην Πρίστινα, δηλαδή ότι το κυρίαρχο κοσυφοπέδιο θα σκεφτεί σοβαρά να συγχωνευτεί με τη μίζωνα Αλβανία. Πάντα έλεγα ότι αυτό είναι παραμύθι για να φοβίζουμε τα παιδιά, αλλά συζητείτε τώρα και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Και φαίνεται ότι αν το σενάριο δεν μπορεί να αποκλειστεί στην ολότητά του, θα επηρεάσει και τη Μακεδονία ή την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία κλπ. Και σίγουρα επηρεάζει τη Σερβία. Και εμείς πρέπει να το δούμε αυτό το σενάριο, να δούμε τη σημασία που μπορεί να έχει στο μέλλον της δημοκρατίας και στο Κωσυφοπαίδιο και στη Σερβία. Σταματώ εδώ και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Η κυρία Κοπά ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ειλικρίνειά του που κατέστησε δυνατή την υποβολή κοινών τροπολογιών για τα κοινά αποτελέσματα στη μάχη κατά της διαφθοράς, για τις σωστές ε, δίκες δίκες και να υπογραμμίσει και την ε, περιφερειακή συνεργασία και τις καλές γειτονικές σχέσεις. Υπάρχουν κάποια ακόμα θέματα που ελπίζω ο να τα βελτιώσει με τις προτάσεις του, τις συμβιβαστικές. Ένα θέμα που πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα είναι η ανάγκη να υπάρχει καλή ισορροπία μεταξύ του ζητήματος του κοσυφοπεδίου και άλλων θεμάτων που αφορούν τη διαδικασία εκδημοκρατισμού ή καλύτερα την ε, εδραίωση της δημοκρατίας στην ίδια τη Σερβία. Όπως είπα, στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση, κατά την επίσκεψή μας ε, στη Σερβία ε, η κοινωνία των πολιτών μας λέει ότι ε, μπορεί να χάσουμε αυτά που ενδιαφέρουν τους πολίτες της Σερβίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει χωριστεί έκθεση για το που θα συζητηθεί σήμερα και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια μάλλον μαζί στην ίδια Ολομέλεια και ε, πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλά θέματα. Το καλό είναι να συμφωνήσουμε επί δύο-τριών παραγράφων για να αναφέρομαι τα σημαντικά και να διατηρηθεί και η ισορροπία της έκθεσης. Σε αυτά τα πλαίσια θα υπογραμμίσω τις μεγάλες μου αμφιβολίες για την δυνατότητα να τεθεί το θέμα του κοσοϊκοσυφοπεδίου σε σχέση με το Σερβικό Σύνταγμα. Γιατί Ποτέ άλλοτε στην ιστορία της διεύρυνσης δεν ζήτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση από οποιαδήποτε υποψήφια χώρα να ξαναδεί τα ε, σύνορα ή τα κυριαρχικά δικαιώματά της. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ε, επιφυλαχθεί και να κρατήσει τη θέση της ως έντιμο διαμεσολαβητή μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινα και να μην συμμετέχει στην ίδια την ε, αντιπαράθεση. Είναι σημαντικό τώρα που υπάρχει και υψηλού επίπεδου διάλογος μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών με την ίδια λογική θέλω να ζητήσω να γίνουν σεβαστές οι συνομιλίες για το όνομα μεταξύ Ελλάδας και Εφηρόμ και που αναφέρονται στην παράγραφο 23 όπως ε, κάνει και ο ο κύριος Χάουιτ και να αναφερθεί το επίσημο όνομα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονία. Τέλος, ε, στα θέματα που αφορούν την έκθεση, καλό θα ήταν να προσέξουμε περισσότερο τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στη Σερβία, την αύξηση της ανεργίας του δημοσίου χρέους, όπως και τις ανάγκες να ε, τύχουν σεβασμού τα κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Miss Brandner. Thank you very much. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γέλκο για το σχέδιο εκθεσής του και για τις τροπολογίες. Νομίζω ότι έχουμε έτσι μια πολύ καλή βάση για συζήτηση. Από την τελευταία εκθεσή που είχαμε για την Σερβία, η χώρα έχει κάνει περισσότερα βήματα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και έχει προχωρήσει και σε μεταρρυθμίσει στο εσωτερικό. Φυσικά μένουν ακόμα πολλά να γίνουν. Θα αναφερθώ σε μερικά από αυτά. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει ένα που είναι πολύ σημαντικό και που ανέφερε ήδη η κυρία Κοπά που έχει να κάνει με το ε, δικαστικό σύστημα, με τη δικαιοσύνη. Εκεί πρέπει να βελτιωθεί αυτό το σύστημα, η αμεροληπτή, ανεξαρτησία, αποτελεσματικότητα δηλαδή του συστήματος αυτού. Και πρέπει να πάρουμε και μαθήματα από τις αποτυχημένες προσπάθειες που έχουν γίνει κατά καιρού και να καταλήξουμε έτσι σε μια δικαιοσύνη που να σέβεται απόλυτα την ανεξαρτησία της αλλά και να λειτουργεί με ταχύτητα. Το δεύτερο θέμα είναι η διαφθορά. Και εδώ πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία και η κυβέρνηση να βρει τρόπο ώστε να υιοθετήσει μια εθνική στρατηγική κατά της διαφθοράς. Η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει επίσης τους ανεξάρτητους θεσμούς να υπάρξει εισαγγελία ειδική για τα θέματα διαφθοράς και να ενισχυθεί ο ρόλος αυτός και όχι να παραγωνιστεί. Επίσης πρέπει να φροντίσουμε για να σταματήσουν οι διακρίσεις σε βάρος ατόμων, ομοφιλόφιλων, λεζιών κλπ. Πρέπει η κυβέρνηση να καταλήξει σε μια στρατηγική ώστε να καταπολεμήσει την ομοφιλοφοβία και να αντιμετωπίσει ομάδες, χούλιγκαν και άλλες που επιτίθενται σε αυτούς. Πάντως οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις μπορούν να ξεκινήσουν. εμπόδια δεν είναι τέτοιο ώστε να μην μπορούν να ξεκινήσουν. Άσε που η έναρξη τέτοιων διαπραγματεύσεων βοηθάει τη χώρα να προχωρήσει πιο αποτελεσματικά στη, στα βήματα που πρέπει να κάνει. Χαίρομαι επίσης ε, πάρα πολύ για τον ε, διάλογο που έχει αρχίσει το Βελιγράδι με τους πολιτικούς ηγέτες. Ευχαριστώ πολύ την Κάθριν Άστον επίσης για τις προσπάθειες που προσωπικά ήδη κατέβαλε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που παραμένει κλειδί πάντως είναι η εφαρμογή των συμφωνιών και περιμένω την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή αυτή. Η κυβέρνηση πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί επίσης για να καταργήσει τις παράλληλες δομές στο βόρειο Κωσυφοπέδιο. Ελπίζουμε επίσης ότι θα υπερισχύσει το πνεύμα συμφιλίωσης. Το ότι μετέφεραν το μνημείο είναι ήδη ένα δείγμα. Θέλω να θαρρύνω επίση τη Σερβία, το Κωσυφοπαίδιο και την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσουν με τον διάλογο και να συμμετέχει σε αυτό και το Κοινοβούλιο και η Κοινωνία των Πολιτών. Αλλιώ δεν θα υπάρχει αξιοπιστία και στήριξη από τον κόσμο και έτσι υπονομεύεται αυτή η διαδικασία. Εμεί ε, κάνουμε έκκληση στην ομιμότητα και τη διαφάνεια. Ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στον επόμενο γύρο συζητήσεων. Τελευταίο κοιόδη συζητητή ο κύριο Τάνοκ. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον κύριο Κάτσιν για την έκθεση προόδου του για τη Σερβία και φυσικά για την ανακοίνωση ότι η Σερβία είχε γίνει επίσημη υποψήφια για προσχώρηση στην Ένωση και θα ήθελα να ξέρω πότε θα, ξεκινήσει, θα ήθελε να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις. Ε, αναφορά που καλωσορίζω στο άρθρο 359. Για τον ποινικό κώδικα είχαμε παρουσιάσεις, μάλλον μου το ανέφερε ένας ε, σερβικής προέλευσης κάτοικος της περιφερειάς μας, του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία εθνικοποιήθηκαν, ε, ε, απαλωτριώθηκαν ε, με βάση αυτή τη διαδικασία που κατά τη γνώμη μου αντιτίθεται σε οποιαδήποτε λογική και μετά το τροποποίησαν λέει αλλά άλλαξαν τη γλώσσα, τη γλώσσα αλλά διατήρησαν αυτή την αρχή με βάση την οποία μπορούς μπορεί το κράτος να ιδιοποιηθεί της, ε, την ιδιωτική περιουσία. Διαφωνώ με τον συνάδελφο Ζόρζ Σάφλιν, τον οποίον σέβομαι ε, ε, όλος ιδιαίτερο ω ακαδημαϊκό, αλλά η ιδέα του να πούμε τι θα βάλει στο σύνταγμά του μια χώρα, όσον αφορά δηλαδή τη δική του κυριαρχία, σύνορα κτλ, είναι παρέμβαση. Και γιατί να πούμε τότε για την Ιρλανδία που ισχυρίζεται ότι, που ισχυριζόταν μάλλον για 30 χρόνια ότι το βρετανικό κομμάτι του νησιού ήταν δικό της. Πρέπει να σεβαστούμε τις ιστορικές ε, προσδοκίες, ή επιδιώξεις των κρατών. Τα σύνορα αλλάζουν λόγω διεθνούς <coughs> φόβου σε σχέση με την αναγνώριση του κωσυφοπέδιου. Βέβαια το μισό του ΟΗΕ ακόμα δεν αναγνωρίζει το κωσυφοπέδιο και το μισό της Ένωσης δεν αναγνωρίζει το κωσυφοπέδιο και άρα θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να υπάρχει ανεξαρτησία ανάμεσα στην αναγνώριση και την παιδαφική κυριότητα σε περίπτωση χωρών των οποίων τα διεθνή σύνορα δεν έχουν ακόμα καθοριστεί. Πολλοί στη Σερβία τώρα θα περίμεναν να υπάρξουν ανταλλαγές, αυτό αναφέρθηκε σε αντάλλαγμα της σταθεροποίησης της περιοχής και της αναγνώρισης του κοσυφοπεδίου. Αλλά δεν πρέπει να έχουμε εμεί εδώ απόλυτες θέσεις, γιατί μπορεί να κατηγορηθούμε για υποκρισία για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την υπόθεση αυτή. Και τέλος... Uh, τέλος, να καλωσορίσουμε τη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στο Μαυροβούνιο και τη Σερβία. Η Σερβία δεν είχε και πολύ όρεξη να αποχωριστεί το Μαυροβούνιο. Ευτυχώ πήγε καλά η ανεξαρτησία και τώρα είναι πολύ θετικό το ότι σε ανώτατο επίπεδο γίνονται ε, επισκέψεις αμοιβέ. Ο κύριος Κούκαν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο εισηγητής μας κάνει πολύ καλή δουλειά. Χαίρομαι επίσης γιατί περισσότερες ε, τροπολογίες πάνε προς παρόμοια κατεύθυνση και δεν θα δυσκολευτεί πολύ, ελπίζω, να καταλήξει σε συμβιβαστικές. Επίσης χαίρομαι διότι περισσότερες τροπολογίες υποστηρίζουν να μπει η ημερομηνία για αρχή των διαπραγματεύσεων για την ένταξη για τη Σερβία όταν θα πληρεί τις ε, κύριες προϋποθέσεις και προτεραιότητες. Η συνέχιση του διαλόγου με το Κωσυφοπέδιο είναι πολύ σημαντικό πράγμα προφανώς. Γενικά η εργασία και τα αποτελέσματα μέχρι τώρα πρέπει να εκτιμηθούν και πρέπει να ζητήσουμε σωστή εφαρμογή των αποτελεσμάτων από τον διάλογο. Η ενημέρωση, η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων είναι επίσης σημαντικές για να καταλάβει. Βέβαια, πολλές φορές η διακριτικότητα βοηθάει την αποτελεσματικότητα των διαπραγματεύσεων, αλλά εδώ το, η κοινή γνώμη και βεβαίως οι βουλευτές πρέπει να ενημερώνονται για το περιεχόμενο και την πορεία του διαλόγου πληρέστερα από ό,τι μέχρι τώρα. Υπογραμμίζω την ανάγκη για περαιτέρω μεταρρυθμίσει στο δικαστικό σώμα που αναφέρεται και στην έκθεση. Νομίζω ότι η Σερβία πρέπει να βελτιώσει περισσότερο την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα του συστήματος, ενισχύοντας την ανεξαρτησία και αμεροληψία. Ε, είναι η ε, ροχοκοκαλιά του συστήματος και ε, το τομέας αυτός και σημαντικό, σημαντική προϋπόθεση για την ένταξη. Εγώ ανησυχώ ε, σε σχέση ε, με τις υποχρεώσεις που ε, ανέλαβε στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Για το άρθρο 359 και τη, έχω υποβάλει την τροπολογία 71 με συναδέλφους όπως την κυρία Πάκτο και κύριο Σέφλιν σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις. Ελπίζω να συμβάλλουμε στην συζήτηση του θέματος αυτού και στην τελική λύση. Πιστεύω ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να κλείσει το ταχύτερο δυνατόν από τη σερβική κυβέρνηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ε, ενδιαφέρεται για το θέμα και θα παρακολουθήσει τις εξελίξεις ε, για την τύχη του άρθρου αυτού. Τέλος, συμμερίζομαι τις απόψεις του εισηγητή για την κατάσταση του Πρεσέβο Θέλη. Ήταν μια αξιολόγηση ισορροπημένη. Δεν βλέπω να υπάρχει ένδειξη αδυναμίας οποιασδήποτε κυβέρνηση να συμμετέχει στο, σε διάλογο με τις εθνικές μειονότητες για να επιτευχθούν αποτελέσματα. Ούτε είναι ένδειξη αδυναμίας μιας εθνικής μειονότητας ε, να απόσχει από την ανάληψη δράσης που σαφώς ε, σκοπό έχει να ε, αυξήσει τις πιέσεις. Να... Ο κύριος Πόσελτε Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον συνάδελφο Κατσίν και εγώ για τη δύσκολη δουλειά που έκανε στο δύσκολο αυτό θέμα. Δεν θα μιλήσω για το κοσυφοπαίδιο γιατί θα τα συζητήσουμε αυτά το απόγευμα. Όμως θέλω να πω κάτι για το Σύνταγμα της Σερβίας. Λέγαμε προηγουμένως ότι ε, στο βαθμό που η Κροατία και το Μαυροβούνιο ε, έχουν σχετικά μικρά ε, διμερεί θέματα και ότι αυτά πρέπει να λυθούν, και μιλήσαμε για ένα σωρό διμερή θέματα που πρέπει να επιληθούν σήμερα. Γιατί η Μακεδονία μάλιστα πριν αρχίσουμε τις διπλωματικές σχέσεις με τη Μακεδονία απαιτήσαμε από τη χώρα και αυτή ήταν η συμβιβαστική λύση του 98 να γράψει στο Σύνταγμα ότι δεν έχει εδαφικές αξιώσεις από τους γείτονες. Και τώρα θέλουμε να δεχτούμε στην περίπτωση της Σερβίας το Σερβικό Σύνταγμα να αναφέρονται ε, θέματα που αφορούν το 20 φοπέδιο, μια χώρα αναγνωρισμένη από 27 κράτη-μέλη δικά μας, από την, ε, τη ΣΥΠΑ και από, σχεδόν από όλους τους γείτονες. Πώς είναι δυνατόν, δεν το καταλαβαίνω. Πρέπει να ζητήσουμε το πρόβλημα αυτό να λυθεί. Δεν ξέρω ακριβώς πότε, αλλά στην πορεία της διαδικασίας προσέγγισης το πρόβλημα πρέπει να λυθεί. Το ξέρουν όλοι. Τα σχετικά αγγελία θέματα που συζητήσαμε σήμερα δεν έχουν σχέση σε σχέση με ε, συνταγματική αξίωση προς ε, μια γειτονική χώρα. Μην χρησιμοποιούμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Το ίδιο ισχύει και για τις μειονότητες και εδώ αναφέρομαι στο πρέσεβο. Όποιος δεν έχει πάει τον συμβουλεύω να πάει να επισκεφθεί το Πρέτσεβο. Απερίγραπτη φτώχεια. Πρέπει να κάνουμε κάτι για την ε, περιοχή του Πρέτσεβο. Πρέπει να κάνουμε κάτι ούτως ώστε να υπάρξει κάποια συνοριακή επικοινωνία με τη Μακεδονία και το Κωσυφοπαίδιο. Είναι τελείως απομονωμένοι οι άνθρωποι σε αυτή την περιοχή και τα δικαιώματα των ε, μειονοτήτων δεν υφίστανται. Και αν συγκρίνουμε με τα δικαιώματα των μειονοτήτων τουλάχιστον στα χαρτιά δεν το λέω αξιολόγικα. Των Σέρβων στο Κωσυφοπαίδιο βλέπουμε ένα τερα... μια πολύ μεγάλη ανισότητα. Εγώ είμαι κατά της αλλαγής των συνόρων, αλλά πιστεύω ότι οι μειονότητες ε, από τις δύο πλευρές πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα. Και όποιος πιστεύει ότι μπορεί να ανοίγει θέματα συνόρων ή μειονοτικά, και να τα προχωρεί τόσο πολύ και να τα κινεί όπως η Μητροβίτσα, πρέπει να ξέρει ότι οι άνθρωποι στο Πρέτσεβο ζητούν με το ίδιο δικαίωμα τα ίδια πράγματα. Και κανείς δεν ασχολείται με το Πρέσεβο. Το λέω καθαρά λοιπόν, εδώ θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας, αλλιώς θα δημιουργηθεί εμπόλεμη επικίνδυνη κατάσταση και οι κάτοικοι του Πρέσεβο ε, έχουν δικαίωμα και να τιμούν τους νεκρούς τους όπως όλοι οι άλλοι. Γιατί και εκείνοι είχαν θύματα από τον εμφύλιο του Μιλόσεβιτς. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κάτσεν για την εκθεσή του. Ο εκδημοκρατισμός της Σερβίας είναι κάτι πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τη χώρα, αλλά για ολόκληρη την περιοχή. Και πιστεύω πως όλοι μας εδώ πιστεύουμε το ίδιο. Ό,τι έχει συμβεί τον τελευταίο αιώνα ξεπερνιέται μόνο εφόσον προχωρήσουμε στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχουμε αυτό είναι να στηρίξουμε την Σερβία στην διαδικασία της προς ε, την Ευρώπη. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες που κάνει η Σερβία και να τη βιέσουμε και περισσότερες μεταρρυθμίσεις και για τα όσα προβλέπει ή όποια ρύθμιση έχουμε κάνει μέχρι τώρα, Πρίστινα κλπ. Τεράστιο ρόλο ε, παίζουν όλα αυτά για τον κρατισμό της χώρας. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν και ξέρουν σε ένα μεγάλο βαθμό ότι και ποιος ε, φταίει για το παρελθόν και αυτό είναι σημαντικό για το μέλλον, προκειμένου δηλαδή η Σερβία να μπορέσει να ε, περάσει στις ευρωπαϊκές αξίες. Η Σερβία λοιπόν για μένα πρέπει όχι μόνο να ανοίξει τα αρχεία της, αλλά επιπλέον πρέπει να επιστρέψει και στην, στα θμήματα της ε, τέος Γιουγκοσλαβίας... Ε, τα κομμάτια των αρχείων αυτών που τις αφορούν. Αυτό λοιπόν πρέπει πρώτα να γίνει και έπειτα το θέμα της μητρικής γλώσσας, το να μπορεί κανείς να μαθαίνει τη μητρική του γλώσσα, να μπορεί να χρησιμοποιεί τα βουλγαρικά δηλαδή, εκεί όπου υπάρχουν ε, άνθρωποι που μιλούν αυτή τη γλώσσα είναι πολύ βασικό. Ο κύριος Πόσελτ επίσης αναφέρθηκε σε αυτό. Τέλος. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάνει μία αξιολόγηση όσον αφορά τη χώρα. Ζητάω λοιπόν να στηρίξουμε τη σταθερότητα, την μακροοικονομική σταθερότητα της χώρας, γιατί δυστυχώς διαπιστώνουμε να υπάρχουν τέτοια προβλήματα και σε άλλες χώρες. Ο κύριος Αλαβράκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, με μεγάλη συμπάθεια βλέπω την, το αίτημα της Σερβίας να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης και χαίρομαι ιδιαίτερα όταν διαπιστώνεται ότι επιτελείται πρόοδος στις βασικές μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες τις οποίες έχει ο κύριος Κασίν πράγματι έκανε μια αντικειμενική έκθεση. Αυτή η έκθεση είναι αντικειμενική. Ε, βεβαίως ως προς το σημείο 23 διαλόγους ε, δεοντολογίας θεωρώ την επιβεβαιωμένη χρήση της ορθής και καθιερωμένης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ονομασίας ε, ΦΥΡΟΜ. Ε, συμμερίζομαι τις απόψεις του κυρίου εισηγητού, του κυρίου Κασίν σχετικά με τα θέματα ε, διαφθοράς, ε, ελλείψεων του δικαστικού συστήματος, δημόσιας διοικήσεως, της ελευθερίας του τύπου ε, και θεωρώ ότι σε αυτά υπάρχει μεγάλο έδαφος να γίνουν περαιτέρω βήματα. διάβασα τελευταία μια έρευνα της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής ακεραιότητας η οποία βρίσκει τη Σερβία στη 16η θέση από τις 143 παγκοσμίως ως προς τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές με μέσο ετήσιο όγκο περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια στην πρώτη δεκαετία αυτού του αιώνα. Νομίζω ότι ε, εκεί πρέπει να γίνουν πολλά βήματα ούτως ώστε να περιοριστεί ε, το θέμα των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών. Χαιρετίζω την παράγραφο 24 για πάταξη των κρατικών και ιδιωτικών μονοπωλίων και για μετάβαση σε μια ανοιχτή οικονομία της αγοράς καθώς αυτό αποτελεί σημαντικό κομμάτι της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν ενέργειες προς την κατεύθυνση της διαφάνειας των εισαγωγικών ροών, ώστε να καταστεί κλάδος ανταγωνιστικός και να αποφευχθεί η υπερτιμολόγηση η οποία αυτή τη στιγμή έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Ακόμα, Υπάρχει ανάγκη για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ως απάντηση στα υψηλά ποσοστά ανεργίας και στις πληθωριστικές πιέσεις, τα νέα μέτρα λιτότητας από μόνα τους δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικά παρά μόνο εάν συνδυαστούν σε μια πολιτική για την ανάπτυξη. Και πάλι συγχαίρω τον κύριο Σιγητή. Ευχαριστώ κύριε Yes. Before giving the floor... Να δώσω το λόγο στον εισηγητή για το κλείσιμο. Σας θυμίζω ότι η ψηφοφορία θα γίνει την 5η στο Στρασβούργο. 7 Φεβρουαρίου. Θυμίζω επίσης ότι το απόγευμα στις 4.30 η κυρία Γκρουμπ Τζεσίκα αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Σερβίας θα έρθει εδώ. Δεν, το πρόφερα καλά. Συγγνώμη. Κύριε Κατσίν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω όμως ότι πρώτα πρέπει να μιλήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν εκπροσωπείται. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Μ' ακούτε, ε, η Κομισιόν εκφράζει την εκτίμησή της για την εξαιρετική δουλειά που έκανε ο εισηγητής όπως πάντοτε. Συμφωνούμε ε, επί των περισσότερων τροπολογιών και περιμένουμε να δούμε και τις συμβιβαστικές τροπολογίες να σας πω ότι μπορούμε να συμμεριστούμε και να συμπεριλάβουμε στο έργο μας τις περισσότερες ανησυχίες σας, γιατί την άλλη εβδομάδα θα πάμε στο Βελιγράδι, όπου έχουμε μόνιμο διάλογο με τις αρχές και θα συζητήσουμε ακριβώς και για τις μεταρρυθμίσεις ε, και το διάλογο με το Κωσυφοπέδιο που είναι η προτεραιότητα αυτού του εξαμήνου για το κράτος δικαίου λοιπόν, τη δημοκρατία, τον κοινοβουλευτισμό και άλλα θέματα. Θα μεταφέρουμε τις ανησυχίες σας γιατί έχουμε υπόψη μας ε, ε, για την έκθεση στα μέσα Απριλίου θα επικεντρωθούμε στα κρίσιμα θέματα για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις ε, ένταξης και να βελτιωθούν, και να, βελτιωθούν οι σχέσεις με το κοσυφοπέδιο είναι σημαντικό. Θα υπάρξει κοινή ανάλυση από την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα είναι συγκεκριμένο το θέμα στην έκθεση. Με αυτή την ευκαιρία θα κάνουμε ενημέρωση σχετικά με τις ε, εξελίξεις στις μεταρρυθμίσεις να είναι και ένα κίνητρο, στενή κίνητρο για την τωρινή, τις τωρινές εργασίες που είναι σε όλα τα επίπεδα και προς όλες τις κατευθύνσεις. Και εντυπωσιάζομαι από τη δυναμική των ε, μεταρρυθμίσεων της νέας κυβέρνησης που ένα μεγάλο κομμάτι του προγράμματος δράσης ε, εφαρμόστηκε και αυτό θα είναι και η βασική συζήτηση με την Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης σήμερα το απόγευμα. Εδώ καταλαβαίνω ότι ε, και οι τροπολογίες και οι συμβιβαστικές που θα προκύψουν ακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις γιατί ε, γίνονται πράγματα σχεδόν κάθε εβδομάδα. Να σημειώσω ειδικότερα κάποια καινούρια θέματα, καινούριε εξελίξεις. Καταρχήν το 234 και το 359 είναι άρθρα που ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί, είναι σχέδιο, ακόμα εξετάζεται το θέμα από το Κοινοβούλιο, μέχρι την Άνοιξη θα το δουν. Φαντάζομαι λοιπόν ότι θα μας αποσταλούν μηνύματα και έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να πούμε τη γνώμη μας. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει ε, θέματα εφαρμογής και σημειώνουμε και τις ανησυχίες των σερβικών αρχών ότι κάποιες από τις έρευνες, ε, τις θεμητές για το 359, ορισμένες ήταν νομότυπες, ε, αυτές δεν πρέπει να παρεμποδιστούν ή να αποδυναμωθούν από τη νομοθετική αλλαγή. Πολλά θέματα αφορούν λοιπόν την εφαρμογή των διατάξεων και υπάρχουν και θέματα πιο μεσοπρόθεσμα που αφορούν τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του μηχανισμού ολόκληρου του ποινικού κώδικα. Γιατί βελτιώνοντας όλο το σύστημα θα μπορέσουν να ε, εργαστούν σωστά ε, και οι εισαγγελικές αρχές. Αυτό είναι σημαντικό και ένα άλλο επίσης αφορά και κάποια ζητήματα που θίγονται στις τροπολογίες. Ίσως θα υπάρξει σύντομα συνάντηση Λίτσα Χάγκερ, οπότε εκεί θα ε, υπάρξουν καινούργια στοιχεία. Επίσης ο νέος διευθυντής ε, της υπηρεσίας ε, για την, κατά της διαφθοράς είναι μια κυρία επαγγελματίας και ορίστηκε χθες και αυτή η ομάδα ε, φιλοξένησε την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης την περασμένη εβδομάδα ε, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η πορεία των εργασιών τους ε, στο μέλλον και τον τελευταίο Δεκέμβρη ε, υπήρξε νόμος καινούριο για τις κρατικές συμβάσεις που ευθυγραμμίζεται με το, τους, με το, το κεκτημένο της Ένωσης. Τώρα θέλουμε βέβαια να κάνουμε μια πλήρη ανάλυση, αλλά εν πολλή ακολούθησαν τα σχόλια που τους δώσαμε. Και αυτό είναι καλό για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Τέλος, για τις μειονότητες, νομίζω ότι οι περισσότερες τροπολογίες έχουν τη σωστή προσέγγιση, δηλαδή να υπάρξει οριζόντια σύσταση για την καλύτερη ε, εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. Καλύτερα να κάνουμε έτσι παρά να εξειδικεύσουμε στη μία ή την άλλη ομάδα. Σημειώνω επίσης ε, ότι οι αρχές γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικότερα το πλαίσιο και έχω πληροφορίες από τον Σέρβο Διευθυντή για τις μειονότητες και τα ανθρώπινα δικαιώματα ότι θα δουν τα θέματα των μειονοτήτων για να γίνει σωστή συζήτηση ώστε το Εθνικό Συμβούλιο Μειονοτήτων να το χρησιμοποιήσουν και επίσης εν ώψη των νέων εκλογών του 2014 που πρέπει να οργανωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και από εδώ λοιπόν αποδεικνύεται ότι οι αρχές γνωρίζουν τις ανησυχίες μας και ο Διευθυντής είπε ότι τώρα αναπτύσσουν και νέα στρατηγική κατά των διακρίσεων. Αυτά είχα να σας πω και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ο κύριος Κατσινίων ολοκληρωθεί η συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, ε, Πρόεδρε εκπρόσωποι των αντιπροσωπιών από τα Δυτικά Βαλκάνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεισφορά σας. Και σας ευχαριστώ για την βοήθειά σας, τη στήριξή σας κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του εγγράφου αυτού. Από ό,τι φαίνεται η Σερβία προχωράει και αλλάζει από μια χώρα προβληματική για τα Δυτικά Βαλτάνια σε μια χώρα κινητήριο δύναμη προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν γίνει τεράστια βήματα μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Τέσσερις συναντήσεις μέσα σε λίγους μήνες είναι ένα ρεκόρ που πρέπει να εκτιμήσουμε, να του δώσουμε την αξία που έχει. Και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα αυτό και για τις άλλες χώρες στην περιοχή. Γιατί όταν υπάρχει πολιτική βούληση, υπάρχει πάντα και ο δρόμος για να προχωρήσουμε. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να εκτιμήσουμε. Βέβαια, εγώ δεν θέλω να περάσω πολύ χρόνο εδώ σε λεπτομέρειες, μια που θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με την κυρία και αργότερα, την αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση, και θα μα ενημερώσει για τι εξελίξει. Ο κύριο Σόπφλιν πάντω, αναφέρθηκε στο Σύνταγμα. Όπω γνωρίζετε όλε οι χώρε προ ένταξη όταν ανοίγουν τα κεφάλαια 23 και 24 πρέπει να αναβαθμίσουν το Σύνταγμά του. Και το ίδιο ισχύει και για τη Σερβία. Δεν θέλω να συζητήσω για τα επιμέρους άρθρα, είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα και δεν θα ήταν σοφό να βιαστούμε και να ανοίξουμε κάποια κεφάλαια. Εγώ πιστεύω ότι η Σερβία οριμάζει όσο περνά ο καιρό. Ιδιαίτερα θέλω εδώ να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη συμφωνία πάνω σε ένα έγγραφο για τις διαπραγματεύσεις, μια γραπτή δήλωση. Τίποτα δεν ε, συμφωνείτε αν ε, δεν συμφωνήσουν όλοι. Ναι, αλλά αυτό δεν πρέπει να σημαίνει, και απορρίφθηκε ευτυχώ, ότι γι' αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται και καμία προσπάθεια. Όσοι το στήριξαν ε, απέτυχαν. Γι' αυτό λοιπόν Θέλω να ευχαριστήσω εκείνους οι οποίοι ε, δέχτηκαν να εκτεθούν, να αντιπαρατεθούν με αυτούς οι οποίοι πίστευαν ότι δεν έπρεπε να προχωρήσει η διαδικασία. Ο κύριος Σέπλιν είπε επίση κάτι για φιάλτες, φόβους, όσον αφορά την αλλαγή συνόρων και όσον αφορά τον αλβανικό πληθυσμό στα Βαλκάνια. Εγώ εδώ δεν θέλω να βασίζομαι σε διαδόσεις. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην πρόοδο έτσι ώστε η Σερβία να μπορέσει να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις όσο γίνεται πιο γρήγορα. Η κυρία Κοπά μου αναφέρθηκε επίσης σε μερικά πράγματα και θέλω να πω εδώ ότι είναι πολύ σημαντικό κατά τη διάρκεια της τέταρτης συνάντησης ανάμεσα στο Τάτσο και Τάτσι να ασχοληθούν με το θέμα των παράλληλων δομών Υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις για τις μέχρι τώρα συζητήσεις. Θα συνεχιστούν πάντως το Φεβρουάριο και νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε πριν γίνει πρόοδος. Πιστεύω ότι και δύο πλευρές θα προσφέρουν τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο για να βρουν διέξοδο από αυτό το τόσο ευαίσθητο θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη αναφέρθηκε σε αυτό που είπε και η κυρία Μπράτνερ για την στρατηγική κατά της διαφθοράς και για την υπηρεσία ε, αν και έχουν δεχτεί ότι είναι σημαντική αυτή η υπηρεσία, υποσχέθηκαν ότι θα την ενισχύσουν, ότι θα υιοθετήσουν νέα νομοθεσία, συνεπώς προχωράνε και εκεί τα πράγματα και θα θεσμοθετηθεί η υπηρεσία αυτή πολύ περισσότερο στο μέλλον από ό,τι κατά το παρελθόν. Να πω τώρα και δύο λόγια για το Βελιγράδι και την ε, πορεία αυτή των ομοφυλόφιλων, την παρέλαση των ομοφυλόφιλων. Δεν έγινε η παρέντα, εγώ ήμουν έτοιμος να συμμετάσχω. Αυτή τη φορά πιστεύω ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Θα γίνει πρώτα στο Μαυροβούνι και πιστεύω ότι εφόσον στηριχτεί εκεί, πιστεύω ότι και η Σερβία θα είναι έτοιμη πολύ περισσότερο να βελτιώσει την κατάσταση όσον αφορά τον πληθυσμό αυτών των ομοφυλόφιλων. Για τον κύριο Τάνοκ και τον κύριο Κούτσου που είπαν για το άρθρο 359. Συνομιλούμε με τον κύριο Βούτιτς, με τον κύριο Σαλάκοβιτς κλπ. Ε, αυτό που είναι πιο σημαντικό τώρα είναι να μην γίνεται κατάχρηση των άρθρων από τους ε, δικαστές, από τους αγγελείς. Ήταν ο μόνος τρόπος έτσι ώστε να καταλήγουν στη φυλακή άνθρωποι και να πιέζονται να πληρώνουν πρόστιμα στους πολιτικούς σχέτες, ή οποιοδήποτε. Αυτό είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε να αναπτύσσεται εδώ μια χώρα τέτοια ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις μαζί μας. Εμείς θα επιμείνουμε σε αυτό. Όπως ε, πάντως λέει και ο Έντουαρτ, συμφωνώ και εγώ, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που έχουν πάει στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου. Το οποίο είναι ένα μήνυμα βέβαια προς την κυβέρνηση της Σερβίας να κάνει κάτι με τη δικαιοσύνη της. Θα υπάρξουν αλλαγές σε λίγες μέρες και πιστεύω ότι θα έχουν θετικές επιπτώσεις στις μελλοντικέ ε, εξελίξεις. Ο κύριος Πόσελ, όσον αφορά τις προκλήσεις και την ε, ερμηνεία του τι είναι εφικτό και τι δεν είναι θα μπορούσα να συμφωνήσω με κάποια μηνύματα που μετέφερε, αλλά η πολιτική του ομάδα, το ΕΛΚ, νομίζω ότι πρέπει να καθίσει τέτα τέτ με την ηγεσία στο Βελιγράδι να συζητήσουν. Δεν είναι θέμα της έκθεσης αυτής. Είναι θέμα μελλοντικών προκλήσεων που θα προχωρήσουν όσο είναι πιο προφανής και ο διάλογος. Σας είπα ότι όλες οι πλευρές οριμάζουν και μπορούν να προσφέρουν πολύ περισσότερα από ό,τι μπορούσε κανείς να φανταστεί στο παρελθόν. Δεν συμφωνώ με την Κέτη Άστον πάντως για το ότι τα πάντα πρέπει να έχουν γίνει μέχρι το Μάρτιο. Εγώ πιστεύω ότι εκείνη θα έπρεπε να συνεχίσει στο μέλλον να είμαστε περισσότερο φιλόδοξοι και να κάνουμε το δικαστικό σύστημα της Σερβίας ε, και τον κόσμο ε, να το βάλουμε μάλλον σε θέση όπου θα βοηθήσουμε εμείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να αλλάξει. Ο κύριος Κοβάτσης επίσης ανέφερε κάποια προβλήματα. Είμαστε μαζί σε μια επίσκεψη στην βουλγαρική μειονότητα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την ε, υποανάπτυξη από την οποία υποφέρουν οι περιοχές αυτές που βρίσκονται στα σύνορα με την Βουλγαρία. Χρειάζεται οικονομική αρρωγή. Αλλά μέσα σε αυτό το θετικό πνεύμα πιστεύω ότι θα βρούμε μια συμβαστική τροπολογία και θα μπορέσουμε έτσι να συμπεριλάβουμε και τις προσδοκίες των Βουλγάρων συναδέρφων όσον αφορά τη χρήση της γλώσσας στην εκπαίδευση και στους θεσμούς τουλάχιστον να γίνεται αυτό πολύ περισσότερο από ό,τι κατά το παρελθόν. Όπως πάντως γνωρίζετε, τα περισσότερα προβλήματα έχουν να κάνουν με την τοπική κοινότητα και η ηγεσία εκεί δεν ε, είναι πολύ ισχυρή, για να το πω έτσι με ευγενικό τρόπο και έτσι δεν βοηθούν πάντα να υπάρξει βελτίωση. Χρειαζόμαστε ηγέτες που να είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν περισσότερα στον πληθυσμό εκεί. Αυτά δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο για τον κύριο Σαλαφράκο. Απλώς πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε συμφωνία επί του συμβιβασμού σύντομα. Και είμαι αρκετά σίγουρος ότι η τελική έκθεση θα υιοθετηθεί με μεγάλη πλειοψηφία. Και έτσι θα ενισχυθεί το μήνυμα που θα στείλουμε όχι μόνο στη Σερβία και στο λαό της Σερβίας και στην ηγεσία της, αλλά πρώτα απ' όλα στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης. Συνεπώς ολοκληρώνω υπογραμμίζοντας για άλλη μια φορά ότι έχουν επιτευχθεί πολύ περισσότερα πράγματα σε ένα χρόνο από ότι την προηγούμενη περίοδο στη Σερβία. Υπήρξε πολύ σκεπτικισμός όταν ανέλαβε η νέα ηγεσία στο Βελιγράδι, αλλά προς το παρόν όλα καλά. Και πρέπει απλώς να κάνουν τη δουλειά τους και εκείνοι και εμείς να τους βοηθήσουμε όσο περισσότερο και όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή και όλους σας.